Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε συνεδρία. Έχουμε λιακάδα στις Βρυξέλλες. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και παράθυρο στην αίθουσα. Ξεκινάμε. Ζητώ από τους βουλευτές να μου πούν κατά πόσο συμφωνούν με την ημερήσια διάταξη της σημερινή και την αυριανή. Ναι, ευχαριστώ. Ας ευθετήσουμε και τα πρακτικά έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεως 25ης και 26ης Απριλίου εγκρίνονται. Πάμε τώρα στι ανακοινώσει της Προέδρου. Θα ξεκινήσω με τα καλά μαντάτα. Ποια είναι τα καλά μαντάτα. Η ακτή του επεκύρωσε το κάθεστος της, Ρο, το, τη σύμβαση της Ρώμης, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και έχουμε 132 κράτη που έχουν επικυρώσει άλλες εξελίξεις συζητήσαμε την κατάσταση στην Τουρκία, τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. We had cases where... Είχαμε σοβαρές περιπτώσεις όπου οι δικηγόροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνελήφθησαν. Το συζητήσαμε στο Στρασβούργο, στην αντιπροσωπεία για την Τουρκία, στο Κοινοβούλιο, το θέμα της ανεξαρτησίας του δικαστικού κλάδου και την υπόθεση εδώ της Πινάρ Σελέκ, που είναι φεμινίστρια, και κοινωνιολόγος η οποία προσπιζόταν ενεργά τα δικαιώματα των ευαλωτών κοινοτήτων και των Κούρδων και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη για τρομοκρατικές πράξεις σύμφωνα με την καταγγελία, με την κατηγορία αυτή η απόφαση μετά από αθώση που έλαβε χώρα τρεις φορές Άρα είναι σαφές ότι υπάρχουν πολιτικοί λόγοι για αυτή την ε, καταδίκη και την υπόθεση. Παρακολουθούμε, όταν λέω εμείς, παρακολουθούμε μέλη της Επιτροπής, αλλά και η Γραμματεία. Και θα δούμε στις συζητήσεις με την ε, Τουρκία ε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Είχαμε το πρώτο δικαστικό πακέτο που θεσπίστηκε στην Τουρκία και θα δούμε πώς θα πώς θα επηρεάσει μάλλον τις σχέσεις μας με την Τουρκία και στην ετήσια έκθεση προόδου για την Τουρκία θα αντικατοπτρίζεται και αυτή, αυτό το πακέτο για, με τα μέτρα για το δικαστικό κλάδο. Την περασμένη φορά στο Στρασβούργο, στην Ολομέλεια, υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΙΕ. Ήταν πλήρε το ψήφισμα που αποτελεί μια καλή βάση για την αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας που θα μεταβεί εις Γενέβη την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Σύνοδο. Ε, συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής μας το θέμα ε, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Προτεραιότητες θα αφορούν τη Συρία, Μιανμάρ, Βιρμανία, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας και το Μαλί και θα είναι πολύ έντονη μάλλον η συζήτηση και θετήσαμε και κατεπήγοντα ψηφίσματα στο Στρασβούργο για την σύλληψη επανασφιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ζιμπάμπουε κυρίως εκείνων που κινούνται στα πλαίσια των ενώσεων ε, πράσπιστων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό ε, δείχνει ότι έχουν περισσότερες ε, περιστάσεις ε, ομοίης βίας της αστυνομίας κατά των ακτιβιστών. Επίση, καταδικάσαμε και την έλλειψη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πρόσφατη συναψή προσωρινή συμφωνία οικονομική συνεργασία με τέσσερι αφρικανικέ χώρε, συμπεριλαμβανομένου και του Τζιμπάμπουε, και ζητάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριλαμβάνεται τι ρήτρε σε μελλοντικέ διαπραγματεύσει για οικονομικέ συμπράξει με τη χώρα. Μετά ε, έχουμε άλλο ψήφισμα στα κατεπήγοντα που αφορούσε τις δολοφονίες και επιθέσεις κατά ιατρικών, ε, ιατρικού προσωπικού στο Πακιστάν. Γιατί δέχτηκαν επίθεση. Διότι είναι στην Ήπεθρο, είναι στη χώρα αυτή, στην Ήπεθρο για να κάνουν εμβόλια πολυμιολίτιδος και οι τρομοκρατικές ομάδες είναι εντελώ ε, αντίθετες σε αυτό τον εμβολιασμό. Καταδικάσαμε αυτές τις δολοφονίες και τις επιθέσεις συζητήσαμε την κυβέρνηση του Πακιστάν να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας για τέτοιους οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα αυτό ε, και το προσωπικό και τελικά είχαμε ένα ψήφισμα για, την, για τον περίφημο ακτιβιστή ε, του λαού, τον κύριο Σομπάθ Σομφών, ο οποίος εξαφανίστηκε ε, το Δεκέμβριο και η κυβέρνηση είπε ότι ξέρει ότι έχει ε, εξαφανιστεί, αλλά διατείνονται ότι είναι ποινική υπόθεση και ζητήσαμε την κυβέρνηση του Λάος να πραγματοποιήσει έρευνε όσον αφορά την εξαφάνιση του ανθρώπου αυτού. Υιοθετήσαμε και δύο εκθέσει στην προηγούμενη Ολομέλεια όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, μία στην Επιτροπή Γιούρη και μία άλλη στην Επιτροπή Απασχόληση. Και θα θυμόσαστε ότι από την Επιτροπή μα, την Επιτροπή Ιντρουά. Ε, συντάξαμε μια γνωμοδότηση που αποβάλαμε και στις δύο επιτροπές και βλέπουμε ότι κάποιες από τις συστάσεις μας έχουν συμπεριληφθεί όμως σε διαφορετικό επίπεδο, διαφορετικό βαθμό. Ευχαριστώ για τον κύριο Γκζιπ, ο οποίος ε, συνέταξε αυτή την γνωμοδότηση. Θετήσαμε και ένα ψήφισμα για την Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου για την επόμενη σύνοδο στον ΟΗΕ που θα εστιαστεί στην βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και υπογραμμίσαμε στο ψήφισμα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την εφαρμογή των συμπεφωνημένων συμπερασμάτων που ελπίζουμε που θα, ε, στα οποία θα καταλήξουμε τον Μάρτιο. Σαν Πρόεδρος ήμουνα σε μια συνεδρίαση το, της Διευθύνσεως Κώστη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Επιστήμη και Τεχνολογία. Ε, ακούσαμε εκεί μια παρουσίαση που αφορούσε ένα πρόγραμμα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μεταρρύθμιση του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ήταν πλήρης η μελέτη και δεν μπορώ παρά να θαρρύνω όλους σας να το διαβάσετε τη μελέτη. Επέκρινα κάποια σημεία ο Μάνφρεν Νόμακ προεδρεύει από το Ινστιτούτο Μπόλτσμαν της Βιέννης και, και να σε πιστήσω την προσοχή και σε ένα εργαστήριο για την διαφθορά στα, και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τέτοιες χώρες που θα διοργανωθεί από την Τρουά σε συνεργασία με το τμήμα διαμόρφωσης πολιτικής στις 28 Φεβρουαρίου το πρωί και θα προεδρεύει η συνάδελφός μας η Άννα Γκόμες ε, επίσης θα είναι η συγγήτρια για μια έκθεσή μας ε, που θα αφορά το θέμα αυτό και τέλος να σας ε, ενημερώσω για δύο συνεδριάσεις, συναντήσεις που είχα χτες και προχτές. Η μία ήταν με τον πρέσβη της Ταϊβάν, διότι την περασμένη φορά στην Τρουά θέσαμε το ζήτημα των έξι εκτελέσεων στην Ταϊβάν Παραβίαση λοιπόν του παγώματος του μορατόριου, το συζητήσαμε το θέμα αυτό. Ο πρεσβευτής είπε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν ε, γίνεται δημόσια συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση για κατάργηση θανατικής ποινή και ότι υπάρχουν αποκλίνουσες ε, απόψεις στην κυβέρνηση, αλλά όσον αφορά το... Λένε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να καταργηθεί η θανατική ποινή η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση έχουν την ίδια άποψη. Σε αυτή την συνάντηση έμαθα ότι η κυβέρνηση της Ταϊβάν εξέδωσε την πρώτη πλήρη έκθεση τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα της και κάλεσε Επιτροπή Διεθνών Εμπειρογνωμών να συζητήσει την κατάσταση. Τους ενθαρρύνω λοιπόν να συνεχίσουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όπως ε, τους είπα είναι πολύ σημαντικό η πολιτική ηγεσία της χώρας να προσπαθήσει να δημιουργήσει περισσότερη ανοιχτή συζήτηση ε, για το, ότι, ε, το πόσο άσκοπο είναι να επιβάλλει τη θανατική ποινή αν θες να καταπολεμήσει τη σοβαρή εγκληματικότητα. Δεν έχει νόημα. Και συναντήθηκα και τον κύριο Αμντούλ ε, Ραμάν Ράσιντ Μπούντσαπ που είναι στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στο Κοινοβούλιο του Μπαχρέιν τον ευχαρίστησα που μας βοήθησε να διοργανίσουμε να πάει με προσωπία το Δεκέμβριο από την Επιτροπή μας στο Μπαχρέιν και σε κάποια ζητήματα γίνεται πρόοδο στο Μπαχρέιν αλλά είναι πολύ αργός ο ρυθμός και πρέπει να υπάρξει διάλογος με την αντιπολίτευση όσον αφορά την εφαρμογή των διαφόρων μέτρων, υπάρχει συνέπεια όσον αφορά της, ε, την έκθεση για την έρευνα για τις ε, ταραχές που είχαν σημειωθεί εκεί. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας καλωσορίζω όλους, αλλά ιδιαίτερος καλωσορίζω δύο συναδέλφους από μη κυβερνικές οργανώσεις από την Καμπότζη. Εργάζονται για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έναν φορέα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα σύνδεσμο και εργάζονται για την κοινότητα, για ένα κέντρο, για την ε, εκπαίδευση, νόμιμη εκπαίδευση, νομική εκπαίδευση και έχουμε ετοιμάσει δύο ψηφίσματα εμείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρέστα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τις ε, εκχωρήσεις ε, γεών και έχουμε και προσωπικό της Διεθνούς Αμνηστίας από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και από Ισραήλ και από την Ισία που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το έργο που γίνεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ευχαριστώ που ήρθατε. Και τώρα θα ασχοληθούμε με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη και έμαθα κάτι το οποίο είναι ατυχές ότι παρόλα τα μέσα που στη διάθεσή μας δεν καταφέραμε να, να φτάσει η επίσημη πρόσκληση στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτελικής ε, Ασίας. Στείλαμε την πρόσκληση όμως. Πρέπει να ερευνήσουμε γιατί δεν κατέφθασε η πρόσκληση, διότι ήρθε ο Πρόεδρος και είναι αδύνατο να παραστεί, να είναι εδώ, διότι θα πρέπει να ε, υπερασπιστεί τη δική του και να παρουσιάσει την εκθεσή του σε άλλη επιτροπή. Τώρα, σαν αφορά τα αλλαγή απόψεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες, στην περιοχή της Ασίας, χώρες Άζια, είμαστε περι... θέλουμε να μάθουμε ως Περιφερειακό Κοινοβούλιο τι κάνουν οι άλλες περιφέρειες για να βελτιώσουν την κατάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή τους. Είχαμε αρκετές συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων με συναδέλφους ε, των κοινοβουλίων και με χώρες της ε, περιοχής Άζεαν συζητήσαμε και πριν υιοθετηθεί η διακήρυξη των χωρών Αζέαν για τα ανθρωπίνα δικαιώματα, πέρσι συζητήσαμε τα θέματα. Οι αρχικοί κρατών κυβερνήσεων θέτησαν το κείμενο των κρατών μελών τη ε, περιοχής ΑΖΕΑΝ. Και βέβαια ήταν καλό και είναι καλό ότι θα υπάρξει με τη διακήρυξη. Αλλά ήδη είδαμε στην σύνταξη, κατά τη σύνταξη αυτού του κειμένου ότι υπάρχουν πολλές επικρίσεις όσον αφορά την διατύπωση. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η συζήτηση δεν έλαβε μόνο χώρα εδώ, στην δική μας την Επιτροπή, αλλά και η Πατή Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρία Πιλάη, παραδέχτηκε ότι είναι πολύ καλό το ότι η περιοχή, η περιφέρεια Άσεν ε, καταβάλει προσπάθειες ούτως ώστε να βελτιώσει την κατάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα και να κάνει το κατάλληλο έργο. Επίσης υπογράμμισε όμως ότι τα, τα, οι προδιαγραφές οι παγκόσμιες τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα καθολικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να είναι βάση και ξέφρασε ανησυχία γιατί οι περιφερειακοί φορείς πρόσφατα υιοθέτησαν αυτή τη διακήρυξη τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, που έχει μια διατύπωση που δεν συνάδει με διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα τούτων λεχθέντων θα ήθελα να παρουσιάσω τους εμπειρογνώμονες έχουμε μαζί μας εδώ να ακούσουμε πρώτα τι έχουν να μας πούν πριν ξεκινήσει η συζήτηση έχουμε την κυρία Ισαμπέλα Αραντών, υποδιευθύντρια του προγράμματος Ασίας Ειρηνικού, προς τα που που είναι, σας ξέρω, ξέρω από τα πρόσωπά σας. Ισαβέλα, ναι, ήσουν μαζί μας από τη Διεθνή Αμνηστία για το πρόγραμμα Ασίας Ειρηνικού, ήσουν μαζί μας όταν ε, συζητήσαμε το κείμενο για τη διακήρυξη των χωρών Ασίαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε και την κυρία Γκαέλ Ντουσεπούλκρε, της Σεπιλκρέ από το FIDH, ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή Άζεαν. Είμαι πολύ ικανοποιημένη και χαρούμενη ε, που έχουμε εκπροσώπους από αρκετές χώρες της περιοχής Άζεαν. Καλώς ήρθατε. Καλωσορίζω ιδιαίτερα τον πρέσβη της Μαλαισίας, τον κύριο Ταρτοτσάιν Λουμπίν. Γεια σας. Πρέπει τώρα να ξέχασα και έψαχνα να τον βρω. Ο κύριος Ρόρι Μαγκόουαν, επικεφαλής του τμήματος Ασίας Ειρηνικού, του τμήματος ε, ε Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, δεν είναι εδώ. αλλάξουμε τη σειρά. Λοιπόν, ακούσουμε πρώτα την κυρία Ραντόνα από τη Διεθνή Αμνηστία. Μπορείτε να ξεκινήσετε με την παρουσίασή σας. Thank ευχαριστώ πολύ για αυτή την φιλική εισαγωγή, ευγενική εισαγωγή και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παραστώ εδώ σήμερα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναξεκινήσουμε να προβληματιζόμαστε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Κάνοντας αυτό ξεκινώ ίσως με την περίπτωση της ε, κοινωνίας των, Σάμπατ, ε, των υπέρμαχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σάμπατ Σονχάν. Έχετε νομίζω υπόψη σας αυτό το μήνα αυτή την περίπτωση. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που πρέπει να θυμόμαστε πρωτού ξεκινήσουμε οτιδήποτε. Είναι πολύ γνωστή η εργασία για την εκπαίδευση, παιδεία, συνειδητοποίηση και μετά από την σύλληψη στο Βιεντιάνε την 15η Δεκεμβρίου 2012 και την, τον τραυματισμό του κανένας δεν τον ξαναείδε από τότε και ο λόγος για τον οποίο θέλω να προβληματιστούμε για αυτή την περίπτωση αυτού του ατόμου είναι επειδή η περίπτωσή του είναι συμβολική για το τι συμβαίνει με υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνολικά στην ε, ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας σήμερα υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Νοτιοανατολική Ασία ενοχλούνται προπυλακίζονται, διώκονται και σε κάποιες περιπτώσεις δολοφονούνται κιόλα ή απάγονται. Υπάρχουν πολλοί ε, αναποτελεσματικά συστήματα δικαιοσύνης και προσαγωγή στην δικαιοσύνη των θητών και των εγκληματιών. Υπάρχει επίσης και απουσία περιφερειακού μηχανισμού ώστε να αποκατασταθεί η τάξη σε αυτό το πλαίσιο και σε σχέση και με την ε, ε, οποιαδήποτε ε, συνέχεια μπορεί να δοθεί σε τέτοιου είδους παράπονα ή προσφυγές για την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να προσέξουμε, θα ήθελα να αναφέρω τρεις τομείς. Ο τομέας της ελευθερίας της έκφρασης, η κατάσταση των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Νοτιοανατολική Ασία, σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη και την ποινή θανάτου που επιβάλλεται. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε πολλές χώρες στην Νοτιοανατολική Ασία όσον αφορά την σύλληψη και κράτηση ειρηνικά διαμαρτυρώμενων διαδηλωτών και πρέπει εδώ πραγματικά να λάβουμε υπόψη το ότι υπάρχει έκδηλη βία όσον αφορά τέτοιου είδους ειρηνικέ διαμαρτυρίες. Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συναθρίζεσθε και υπάρχουν αυτά τα εγκλήματα εις βάρος των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς να τιμωρούνται υπεύθυνοι. Στο Βιετνάμ, στο 2012, δεκάδες άτομα βρέθηκαν στις φυλακές με μεγάλες ποινές φυλάκισης ε, που δεν ε, τηρούν με κανένα τρόπο τις διεθνείς προδιαγραφές. Ε, το Σεπτέμβριο 2012, για παράδειγμα, τρεις bloggers μαζί με τον Γκουγέν Φανχάν προσήχθησα στα δικαστήρια διότι έκαναν λέει προπαγάνδα κατά της ε, ε, καθεστικίας τάξης, κατά της κυβέρνησης. Επίσης ε, οι ιδρυτές της λέσχης δημοσιογράφων έτυχαν της ίδιας αντιμετώπισης. Εξακολουθεί να απουσιάζει η ελευθερία της έκφρασης και φέτος στις 9 Ιανουαρίου 2013 ήδη 13 ειρηνικοί διαδηλωτές καταδικάστηκαν μεταξύ τριών και 10 ετών φυλάκισης γιατί έκαναν λέει δραστηριότητες για την ανατροπή της κυβέρνησης του Βιετνάμ. Οι αρχές της, του Βιετνάμ υποψιάζονται ότι υπάρχουν εδώ πολιτικές διασυνδέσεις που θεωρούνται ύποπτες. Ε, εδώ ε, ο ισχυρισμός είναι ότι υπάρχουν και διασυνδέσεις με ε, τρομοκρατικές οργανώσεις για την Καμπότζη. Στο ψήφισμα αναφέρονται οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με την Καμπότζη. Μέλη της ε, κοινότητας ε, των υπέρμαχων ανθρωπίνων δικαιωμάτων διώκονται, προπυλακίζονται, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του 2012. Ας αναφερθώ στην περίπτωση Μαν 70 71 που είναι ε, ε, έγκριτος δημοσιογράφος και που έχει ε, πολύ γνωστή δουλειά που έχει αναπτύξει μέσω τέτοιων σταθμών η κατηγορία είναι ακριβώς ότι έκανε αυτές τις δραστηριότητες υπέρ της δημοκρατίας. Έχουμε επίσης και την κατηγορία που επιβάλλει τις βαρύτερες ποινές με καταδίκη 20 ετούς φυλάκισης τον Οκτώβριο 2012. 20 ετούς φυλάκισης. Και βλέπουμε εδώ επίσης και σε σχέση με τα όσα προβλέπονται για το Μάρτιο 2013 προ ε, σας προσκαλώ να ε, παρατηρήσετε προσεκτικά το τι θα συμβεί τον Μάρτιο 2013 σε σχέση και με την ε, προσφυγή για το ότι η δίκη αυτή δεν ήταν δίκαια. Τώρα σε σχέση με την διεκδίκηση δικαιωμάτων στέγασης στην Καμπότζη αντιμετωπίζουν υπέρμαχοι δικαιωμάτων όλο και αυξανόμενη βία το 2011. Είχαμε και τον, ε, ε, τη δολοφονία ε, ατόμου σε μια επαρχία, καθώς επίσης και την εκδίωξη 600 οικογενειών. Ένας συνδικαλιστής προπυλακίστηκε και οδηγήθηκε στα, στα κρατητήρια τον Ιούλιο πέρυσι. Δεν έγιναν επαρκείς διακριβώσεις για το τι συνέβη με αυτούς τους πολίτες. Ταϊλάνδη τώρα. Η ελευθερία της έκφρασης εξακολουθεί να ε, περιστέλλεται λόγω της ε, νομοθεσίας ε, που υφίσταται σε σχέση με το βασίλειο αυτό με βαρύτατες πηγές φυλάκισης όσον αφορά για παράδειγμα προσβολή της μοναρχίας ως θεσμού. Εφέτος στις 23 Ιανουαρίου 2013 είχαμε καταδίκη σε δεκαετή φυλάκιση διότι δημοσιεύθηκαν άρθρα τα οποία υποτίθεται ότι θίγουν το θεσμό της ε, Βασιλείας. Η Διεθνής Αμνηστία θεωρεί ότι είναι κρατούμενο συνείδησης ε, ο δημοσιογράφος αυτός. Μαλαισία τώρα σε σχέση με την κατάσταση που αντιμετωπίζουν ε, όσοι ασκούν επικρίσεις ε, στις αρχές και στην κυβέρνηση και διεκδικούν δικαιώματα για τις ε, λεσβίες και τους ομοφιλόφιλους διώκονται και τιμωρούνται αυστηρά. Εξακολουθούν να υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις που περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης ως δικαίωμα. Ινδονησία. Η Διεθνή Αμνησία έχει τεκμηριώσει δεκάδε συλλήψεων όσον αφορά ειρηνικέ ε, διαμαρτυρίες ε, υπέρμαχων των ε, δραστηρίων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποιοι από αυτούς καταδικάστηκαν σε μακρότατες ποινές φυλάκισης, από τριετή φυλάκιση μέχρι εικοσαετή φυλάκιση. Ένας δάσκαλος έχει υποστεί ποινή φυλάκισης 15 ετούς διάρκειας ε, διότι άσκησε επικρίσεις σε σχέση με τον πρόεδρο Μπαμπόγκ και σε σχέση με την ε, ε, σημαία που ανατήθηκε για την ανεξαρτησία μιας περιοχής της Ινδονησίας. Βρίσκονται πάρα πολύ στις φυλακές της Ιάβας, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις οικογένειές τους. Επίσης, χρησιμοποιείται νομοθεσία για να καταδικάζονται σε ποινέ φυλάκιση ε, υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απλά επειδή διεκδικούν τα δικαιώματα να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους δικαιώματα και να εκφράζονται ελεύθερα. Και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το καθεστώς καταστολής. Τον Ιούλιο 2012 Μούλουκ από την Ανατολική Ιάβα καταδικάστηκε για βλασφήμια σε διετή ποινή φυλάκησης ο ειδικό ε, εκπρόσωπος ε, ε, αντεταλμένο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προσέλθει στην Ινδονησία για να διακριβώσει το τι συμβαίνει. Δεν έχει καθοριστεί όμως η ημερομηνία. Ευελπιστούμε ότι ο ειδικό απεσταλμένος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορέσει να επισκεφθεί αυτή την χώρα και να διακριβώσει το τι γίνεται. Υπάρχουν επίσης παραβιάσεις ε, των ε, δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών των ε, ατόμων που παραμένουν όλες αυτές οι περιπτώσεις χωρίς να έχουν επιληθεί. Έχουμε και την δολοφονία Μουνία Σάκερ Κάλεκ που όλα αυτά τα οποία συναρτώνται με την δολοφονία αυτή δεν έχουν διακριβωθεί με κανένα τρόπο μέχρι σήμερα. Φιλιππίνες. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ε, το θέμα της ατιμορρησίας δολοφόνων ε, δημοσιογράφων στο ε, Μιντανάο. Από τη σφαγή στο Μιντανάο τόσο καιρό πέρασε και διασφάλισαν οι αρχές των Φιλιππίνων ότι θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Από το Σεπτέμβριο 2009 από τους 197 από, από τους 197 υπόπτους ε, οι περισσότεροι είναι ελεύθεροι. Δεν υπήρξε καμία μορφή δίωξης εις βάρος τους. Και εδώ έχουμε και περαιτέρω ε, βιοπραγίες και δολοφονίες σε σχέση με τις ε, οικογένειες αυτές των θυμάτων. Μιανμάρ, Βιρμανία Δεν θα επισέλθω σε πολλές λεπτομέρειες για τη Μιανμάρ, γιατί θα έχετε μια ξεχωριστή συνεδρίαση που θα αφιερωθεί στην περίπτωση της Μιανμάρ. Υπάρχει κάποια πρόοδος που έχει σημειωθεί, όμως υπάρχουν ε, περιοριστικές νομοθετικές διατάξεις για την ελευθερία της έκφρασης, ε, καθώς επίσης ε, και παρά την απόφαση να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, εξακολουθούν να βρίσκονται στα κρατητήρια πολλοί από αυτούς με ευχαρίστηση θα σας διαθέσουμε περισσότερα στοιχεία όταν θα έρθει η ώρα να εξεταστεί το θέμα της Μιανμάρ. Αυτοί οι περιορισμοί στην ελευθερία της εκφρασής ε, πρέπει να εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο μιας αποδυναμωμένης ε, δικαστικής τάξης πραγμάτων. Και πρέπει να θυμάται κανείς ότι σε πολλές από αυτές τις νοτιοανατολικές χώρες Μιανμάρ, Ινδονησία, Καμπότζη υπάρχει ένα κληροδότημα παραβίασης, ε, παράδοση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτά πρέπει να αποκατασταθούν και να τεθεί σε τάξη το σύστημα στην Καμπόζη για τις διακριβώσεις ε, για το τι συνέβη σε σχέση με το καθεστώς των Ερυθρών Κμέρ με πολύ βραδείς ρυθμούς προχωρούν τα πράγματα πέντε άτομα που είναι ύποπτοι για πράξεις γενοκτονίας ε, οι διακριβώσεις δεν έχουν προχωρήσει καθόλου και σε σχέση με την Ινδονησία προφανώς δεν έχει υπάρξει πρόοδος σημαντική όσον αφορά την προσαγωγή εγκληματιών προηγούμενων παλαιότερων εγκλημάτων όπως για παράδειγμα στο Ανατολικό Τιμόρ δεν υπάρχουν εκεί δεν υπάρχει συνεργασία σε σχέση με την έκδοση και παράδοση ε, τέτοιου είδους ατόμων. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν ε, διαπράξει τέτοια εγκλήματα και κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. Αυτή η κατάσταση έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του συστήματος ποινική δικαιοσύνης. Αν δεν μπορέσει να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη σε σχέση με αυτά τα εγκλήματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι αξιόπιστα αυτά τα συστήματα και η έννοια του κράτους δικαίου. Στρεφόμενοι στο κράτος δικαίου όσον αφορά την ποινική δικαιοσύνη σήμερα, η Διεθνής Αμνηστία εξετάζοντας τα όσα τεκταίνονται σε σχέση με την ελευθερία της έκφρασης και αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβαίνουν πολλά και υπάρχουν πολλές ε, λήψεις και παρακολουθούμε τα πράγματα εκ του Έχουμε βασανιστήρια και ε, βιοπραγίες εις βάρος ε, κρατουμένων προκειμένου να υπογράψουν κάποιες ομολογίες. Επίσης η απουσία επαρκούς νομοθεσίας, επαρκούς ισχυρής νομοθεσίας ώστε να ε, μπορούν να καταδικάζονται τέτοιου είδους πράξεις ε, βασανιστήριων. Δεν υπάρχουν πολλές φορές οι αποτελεσματικοί ορισμοί, π.χ. στην Ινδονησία, παρότι υπάρχουν στοιχεία για τέτοιου είδους βασανιστήρια μέχρι σήμερα, οι ορισμοί στον ποινικό κώδικα δεν ανταποκρίνονται, δεν μπορούν να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων σε σχέση με τις διεθνείς προδιαγραφές για την αντιμετώπιση του προβλήματος των βασανιστήριων και των ε, βιοπραγιών κατά των κρατουμένων. Ιδιαίτερα όταν έχουμε περιπτώσεις ε, ειρηνικά ε, διαδηλωτών που ειρηνικά διαδηλώνουν στη χώρα αυτή. Θα πρέπει το πρόβλημα των βασανιστήριων και των, ε, της εξαφάνισης πολιτών οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Εξακολουθούν και υποβάλλονται στοιχεία για τέτοιου είδους εξαφανίσεις και παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όμως είναι τόσο βραδύς ο ρυθμός ε, συμμόρφωσης και επιβολής του κράτους δικαίου που υπάρχει τεράστιο χάσμα, τεράστιο κενό προκειμένου να αποκατασταθούν τα δικαιώματα των θυμάτων στην καθημερινή πρακτική. όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης και των δικαιωμάτων των πολιτών με ε, τα συστήματα τα οποία λειτουργούν στην Νοτιοανατολική Ασία και πάλι εδώ για την Μίανμα ξεχωριστή αναφορά λόγω των τεράστιων προβλημάτων που υφίστανται εκεί. Είναι μια περιοχή αυτή όπου η θανατική ποινή εξακολουθεί να ε, υφίσταται και υπάρχει ευρύτερη συνένεση από πλευράς της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργηθεί αυτή η κατάσταση. Εξακολουθούν να, ε, εξακολουθούν να επιβάλλονται θανατικές ποινές σε πολλές από αυτές τις χώρες στο Βιετνάμ σε σχέση με τις ε, θανατηφόρες ενέσεις ε, που γινόντουσαν για την ε, επιβολή της θανατικής ποινής πάρα πολλοί περιμένουν στα κελιά τους την στιγμή της εκτέλεσής τους. Το ίδιο και σε σχέση και με την Ινδονησία. Υπήρχαν κάποιες θετικές κινήσεις ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των, της θανατικής ποινής αλλά ελπίζει η ε, Διεθνής Αμνηστία ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις σε σχέση με τις χώρες όπου άνομες δίκες ε, λαμβάνουν χώρα είναι ακόμα πιο ανησυχητικό να βλέπει κανείς ότι εξακολουθεί να υπάρχει θανατική ποινή ε, ως ίστατο ενδεχόμενο και μας ανησυχεί αυτό ιδιαίτερα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σε σχέση με ε, την κατάσταση στο περιφερειακό επίπεδο όπως προανέφερα το περιφερειακό αυτό πλαίσιο θα πρέπει να ε, θεωρήσουμε ότι δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα όσα έχουν σήμερα. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα για να διασφαλιστεί ότι θα αποκατασταθεί η κατάσταση πραγμάτων στο μέλλον δεν είναι δυνατόν να συγκρίνει κανείς ε, την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την Ευρώπη και το ασιατικό πρότυπο. Η δήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διακήρυξη για τα, δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες ΑΣΕΑΝ είναι αποδυναμωμένη και δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε ότι αυτή μπορεί να καλύψει επαρκώς ε, το θέμα αυτό επαναλαμβάνομαι στο πλαίσιο της ε, προσπάθειας ε, για την ε, δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου που λέει ως διακήρυξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέσει στο επίκεντρο των προσπαθειών της τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει το Ευρωκοινοβούλιο ρόλο σπουδαιότατο να διαδραματίσει για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που συμβαίνουν και λαμβάνουν χώρα σήμερα στην ανατολική Ασία ζητούμε, απευθύνουμε έκκληση συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει την δημιουργία και εγκαθίδρυση συστημάτων ποινική δικαιοσύνης για την προσαγωγή στην δικαιοσύνη των εγκληματιών. Να υπάρχει η, η δυνατότητα να προχωρήσουμε και να προσπαθήσουμε να προστατέψουμε την ελευθερία της έκφρασης και τα δικαιώματα του ανθρώπου και να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες για την κατάργηση της θανατικής ποινής και να υποστηρίξουμε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται διεθνώς κατά της θανατικής ποινής. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστούμε πολύ. Και θα δώσω το λόγο τώρα στην Γκαέλ από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. <coughs> Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα κάνω την παρέμβασή μου στα γαλλικά. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μιλήσω για την κατάσταση σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Θα ξεκινήσω με το θέμα των διωγμών και της δίμευσης γεών στην Καμπότζη και στην Βυρμανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει κάποιες εγγυήσεις για αυτό το θέμα όσον αφορά την χορήγηση ή τη διατήρηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ε, και ε, εδώ στην Επιτροπή Ιντρουά είναι σημαντικό αυτό το θέμα, ιδίω αν ληφθούν υπόψη τα μέτρα που λήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2012, που αφορούν το, την ανάγκη να διατηρήσουμε το θέμα αυτό μέσα σε όλες τις πολιτικές το θέμα δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να εντάσσεται σε όλα τα θέματα και στις εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η δική μας Ομοσπονδία πιστεύει ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, ε, για συγκεκριμένες ε, υποθέσεις ε, στο Βιετνάμ, στην Καμπότζη και στο Λάος, θα πω δύο λόγια επίσης. Και θα μιλήσω λίγο και για την Ινδονησία και τις τελευταίες εξελίξεις. Ξεκινώ λοιπόν με την Καμπότζη. Υπάρχουν εκπρόσωποι τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως είπε η κυρία Λόχμπιλντερ. Επομένως, μπορείτε να κάνετε ε, άμεσα ερωτήσεις στους παρευρισκομένους από αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αν θέλετε να μάθετε κάτι για τις λεπτομέρειες. Ο κύριος Βίρα Ντεκλέκ και η κυρία Εύη Σούλερ Τελικαντό που είναι ε, μια οργάνωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λοιπόν, σχετικά με την Καμπότζη θα ήθελα να χαιρετήσω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου του 2012 που περιγράφει πολύ καλά την κατάσταση ε, της δίμευσης γεών και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με αυτή τη δίμευση γεών. Παράνομη κράτηση, καταπίεση, ακόμη και ε, δολοφονίες ε, διαφωνούντων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει επιτόπου μια έρευνα για τις σημαντικές αυτές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του κανονισμού για τις εμπορικές ε, προτιμήσεις, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Η Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θέλει να δώσει κάποιες ε, διευκρινήσει ε, για όσα έχουν γίνει μετά το ψήφισμα του Οκτωβρίου 2012 και για τις προοπτικές που υπάρχουν από εδώ και πέρα. Καταρχήν, να σα πω για τι τελευταίε εξελίξει. Οι οικονομικές ε, παραχωρήσεις γεών γίνονται από την κυβέρνηση της Καμπότζης, γνωρίζοντας ότι το Μάιο του 2012 έγινε ένα μορατόριο. Δυστυχώς υπάρχουν κάποια κενά στην οδηγία και δεν υπάρχει και διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία αυτή και συνεχίζουν να δίδονται τέτοιες παραχωρήσεις ε, γης. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αναφέρει 12 τέτοιου είδους παραχωρήσεις γεών. Τώρα υπάρχουν 15 τέτοιες παραχωρήσεις ε, που σημαίνει πάνω από 90.000 εκτάρια που παραχωρήθηκαν μετά ε, το μορατόριο. Το δεύτερο πρόβλημα έχει σχέση με την καταπίεση και την καταστολή των διαμαρτυριών που γίνονται γύρω από, από αυτό το πρόβλημα της δίμευσης γεών και ούτε και σε αυτό το θέμα είναι καλή η κατάσταση. Από τον Οκτώβριο και μετά υπάρχουν σχετικές αρνητικές εξελίξεις. Έχουν αναφερθεί πολλά σχετικά περιστατικά το Νοέμβριο. Οκτώ χωρικοί κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πνόμπενχ συνελήφθησαν και ε, κρατήθηκαν γιατί ε, είχαν βάλει πάνω ε, στην στέγη του σπιτιού τους ε, ένα πανό που έγραφε SOS μαζί με τη φωτογραφία του Μπαράκ Ομπάμα που θα επισκεπτόταν την Πνομπένχ. Το Δεκέμβριο, στις 13 Δεκεμβρίου, ο κύριος Σονάντο δεν μπόρεσε να απελευθερωθεί εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσής του είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 20 ετών και η ε, έθεσή του θα εκδικαστεί στις 5 Μαρτίου στις 5 η ώρα το πρωί. Ζητάμε λοιπόν από την Διεθνή ε, Αμνηστία να είναι σε εγρήγορση για να παρακολουθεί την εκδίκαση της ε, έφεσης που έχει ασκήσει. Στις 27 Δεκεμβρίου καταδικάστηκε ο Γιον Μπόμφα σε τρία έτη φυλάκισης πάλι στην Πνομπένχα και ε, υπάρχουν συνολικά 12 ε, μέλη της οργάνωσης Λικάντο που είναι η τοπική μη κυβερνητική οργάνωση που έχουμε στην Καμπόζη για τέτοια θέματα. Τώρα, όσον αφορά την παρακολούθηση αυτής της υπόθεσης, ε, δεν έχουμε λάβει επίσημη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προθέσεις της, αν δηλαδή προτίθεται να κάνει κάποια έρευνα για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του Οκτωβρίου. Στις διμερείς μας συζητήσεις, από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ακούσει ποικίλα επιχειρήματα σχετικά με αυτή την έρευνα. Αμφισβητείται η ανάγκη μιας τέτοιας έρευνας. Μας είπαν ότι καταρχήν πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός διεθνούς προστασίας και από τον Οκτώβριο του 2012 υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός γιατί ο ειδικό επεσταλμένος των Εθνών για την κατάσταση στην Καμπότζη έχει τεκμηριώσει τις παραβιάσεις σε σχέση με την δίμευση γεών. Αναφέρονται ως σοβαρές και γενικευμένες παραβιάσεις. Άρα καλύπτονται αυτά τα οποία ζητεί ο κανονισμό για τι γενικευμένε προτιμήσει όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δεύτερο επιχείρημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι μια αναστολή των εμπορικών δικαιωμάτων θα δημιουργούσε τεράστιε δυσκολίε για τον τοπικό πληθυσμό. Οι άνθρωποι επιτόπου δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση, εκδιώκονται από τη γη τους, επομένως ε, έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης ε, και πενιχρέ απολαβές. Πρέπει να επιμείνουμε ε, στο ότι το να γίνουν έρευνες στο πλαίσιο του κανονισμού για τις γενικευμένες προτιμήσεις δεν απαιτεί αναστολή αυτών των προτιμήσεων, διότι η έρευνα θα έχει ως αντικείμενο μόνο το άνοιγμα μιας μακράς περίοδου διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση της Καμπότζης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτύχει συγκεκριμένες πρόοδους επιτόπου. Αυτή η περίοδος διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να κρατήσει και δύο χρόνια με βάση τον κανονισμό που ισχύει τώρα. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίζει να εξετάζει αυτό το θέμα, ούτω ώστε το ψήφισμα του Οκτωβρίου να μην μείνει νεκρό γράμμα, να πιέσετε, αν είναι δυνατόν, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει τις σχετικές έρευνες. Είχε διαπιστωθεί ότι ήταν αρκετά σοβαρή η υπόθεση για να ε, ζητηθεί η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει βέβαια να συμφωνεί το Κοινοβούλιο. Εάν ε, γίνει κάποια διερευνητική αποστολή επιτόπου, η Διεθνής ε, Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιμένει ότι μια τέτοια επίσκεψη, μια τέτοια αποστολή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει επαφές με τα κατάλληλα άτομα, με την κοινωνία των πολιτών δηλαδή και τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών. Συνεχίζω τώρα με την κατάσταση στη Βυρμανία. Η κατάσταση όσον αφορά την δίμευση γεών και τους εκδιωγμούς των πολιτών είναι επίσης πολύ ανησυχητική. Αυτές οι παραβιάσεις επίσης έχουν τεκμηριωθεί από τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση στη Βυρμανία στην έκθεσή του από το Μάιο του 2012 και σε μία άλλη έκθεση του Σεπτεμβρίου του 2012. Ε, παραθέτει τις συγκεκριμένε παραβιάσεις ε, λόγω δίμευσης γιών και λόγω καταστολής των διαμαρτυριών. Η Διεθνής Ομοσπονδία ε, έκανε μια αποστολή επιτόπου που έληξε πριν από οκτώ μέρες και φαίνεται ότι οι ομάδες από την κοινωνία των πολιτών αναφέρουν ότι ολόκληρες κοινότητες και αγρότες εκδιώχθηκαν από τη γη τους και υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα υποδομών. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι ε, φαίνεται ότι επιδεινώνεται η κατάσταση όσον αφορά τις επενδύσεις ε, που γίνονται ή που προγραμματίζονται. Και αυτό το τονίζει και ο ειδικό απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών στην έκθεσή του στην παράγραφο 39. Τονίζεται εκεί ότι η αύξηση των επενδύσεων και το ενδεχόμενο κύμα ιδιωτικοποιήσεων και οικονομικές εξελίξεις στη Βυρμανία ενδέχεται να επιδεινώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στη χώρα. Άρα υπάρχουν κάποιες προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν, κάποια σημεία τονίζονται από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΕ. Επίσης, ο εισηγητής David Martin αναφέρθηκε με συγκεκριμένες συστάσεις και ξέρετε ότι υπάρχει ε, ένα σχετικό ψήφισμα στο Κοινοβούλιο που θα συζητηθεί αύριο στην Επιτροπή Ίντα. και αυτές οι προφυλάξεις αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο για την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Ποικίλες προφυλάξεις. Το πρώτο σημείο που τονίζεται από τον ειδικό απεσταλμένο είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ε, για ένα νομικό καθεστώς που θα δημιουργεί ασφάλεια για το καθεστώς ε, ιδιοκτησίας γεών το δεύτερο είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη και πιο συγκεκριμένα για την Μιανμάρ. Θα πρέπει να υπάρξει ένα δεσμευτικό τέτοιο πλαίσιο. υπάρχουν διάφορες προφυλάξεις που πρέπει να λυθούν και θα πρέπει να ε, αξιολογηθούν οι επιπτώσεις και να ελαχιστοποιηθούν ε, οι επιπτώσεις αυτές με παρακολούθηση αυτών των ε, μηχανισμών που θα πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμό επίλυσης διαφορών και υποβολής καταγγελιών. Πρέπει να δοθούν λοιπόν αυτές οι εγγύησει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει κάποια διασφάλιση πριν προχωρήσει περισσότερο στο θέμα αυτό και θα πρέπει να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι για να παρακολουθείτε η κατάσταση και η υλοποίηση των μηχανισμών αυτών με αποτελεσματικό τρόπο. Θα προσπαθήσω να συντομεύσω την υπόλοιπη παρέμβασή μου. Όσον αφορά την ελευθερία έκφραση, ξέρετε ότι η Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε την έκθεσή τη πριν από μια εβδομάδα για την ελευθερία έκφραση στο Βιετνάμ και για την κατάσταση των bloggers. Η Διεθνής Αμνηστία ε, παραθέτει κάποια σημεία ανησυχίας. Δεν θα επανέλθω. Υπάρχει ένα σχέδιο διατάγματος το οποίο θα πρέπει ε, να παρακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, το θέμα αυτό συνδέεται και με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ. Καταρχήν θα πρέπει να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις γιατί η μελέτη επιπτώσεων ε, έγινε το 2008 και δεν λαμβάνει υπόψη τα όσα έχουν γίνει το 2012 όπου έχουμε αποφασίσει ότι θα πρέπει το σύνολο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να περιλαμβάνεται στην αξιολόγηση επιπτώσεων. Θα πρέπει περισσότερο να εξεταστεί ε, λοιπόν το θέμα της ελευθερίας έκφρασης για την κοινωνία των πολιτών και όσον αφορά αυτή τη συνθήκη ελευθέρων συναλλαγών υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο για τους μηχανισμούς παρακολούθησης που προβλέπονται σε αυτή τη συνθήκη θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί παρακολούθησης από την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο του κεφαλαίου για την αηφόρο ανάπτυξη. Και είναι σημαντικό η ελευθερία της έκφρασης ε, να αναφέρεται ρητά, διότι τέτοιο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον παρέχονται κάποιες εγγύησεις. Για την Ταϊλάνδη, Θέλω να τονίσω τη σημασία της υπόθεσης ε, Σομιότ και τη δολοφονία δύο μελών ε, της Ομοσπονδίας Αγροτών από τον Νότο της Ταϊλάνδης το 2012. Και για το ΛΑΟΣ η υπόθεση των σομφών θα πρέπει να παραμείνει στο προσκήνιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος για την ε, Ινδονησία, για τις τελευταίες εξελίξεις θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει ένα νέο νόμο που ονομάζεται ε, προεδρικές ε, οδηγίες ε, υπαριθμών 2 του 2013, διότι αυτό το προεδρικό διάταγμα δεν προσφέρει επαρκείς εγγύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενδέχεται να ποινικοποιούνται ακόμη περισσότερο οι ειρηνικές διαδηλώσεις. Περισσότερε λεπτομέρειε μπορώ να σα δώσω αργότερα, αν θέλετε. Από τον Ιανουάριο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί 18 υποθέσεις βία κατά μειονοτήτων και υπάρχουν και αρκετές υποθέσεις ε, υπάρχουν αρκετά θύματα ε, ε, νεκροί στα πλαίσια κάποιων τρομοκρατικών ε, ερευνών. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μαγκόβεν, θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρεσβευτή του Μπρουνέη, την εξοχότητά του, του συμπίνει Άλλη, Καλώς ήρθατε. Έχουμε και εκπροσώπους από την πρεσβεία της Ταϊλάνδης, της Ινδονησίας, των Φιλιππινών και της Ινδονησίας. Ευχαριστώ όλους σας. Καλωσορίζω, όρισα τον πρεσβευτή της Μαλαισίας ήδη. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Είναι πολύ ευπρόσδεκτο. Με κάποιους από εσά είχαμε και πολύ ε, ενδιαφέρον συζητήσει κατά το γεύμα πριν από μερικούς μήνες. Διότι υπήρχε εντύπωση ότι συνεχώς επικρίνουμε και ότι δεν σημειώναμε και τις θετικές εξελίξεις της χώρας σας. Κατάλαβα την άποψή σας, ελπίζω να κατανοήσατε τη δική μας. Βασικό καθήκον της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι να εστιάζεται επί θεμάτων που είναι προβληματικά. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και οι δύο σας θέσα τα θέματα για το Μιανμάρ ότι στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων στις 4, μάλλον στις 5 Μαρτίου ο πρόεδρος της Μιανμάρ ε, θα παρίσταται και η εδώ πρεσβεία προετοιμάζει πυρετοδό στην εκδήλωση αυτή. Και ίσως θα μπορούσε να συμπεριλάβουμε αυτά που είπατε ε, στη συζήτηση που θα λάβει η χώρα στην ΑΦΕΤ. Ο κύριος Ζόρι Μαγκόβεν επικεφαλής του τμήματος Ασίας Ειρηνικού του ΣΥΠΑ της Αρμοστίας του για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Έχουμε άριστες σχέσεις συνεργασίας με το γραφείο σας των Βρυξελών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέσβεις, εξοχότητες, από τις αποστολές Άζεων και συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω να κινηθώ προς την κατεύθυνση που αναφέρατε κυρία Πρόεδρε, με ισορροπημένο τρόπο να παρουσιάσω επιτέγματα και πρόοδου στην περιοχή, στο χώρο ΑΖΕΝ και κάποια από τα εφιστάμενα προβλήματα, προκλήσεις. Ε, λίγα λόγια να πω όσον αφορά το έργο της ε, του γραφείου του είπατε εκπροσώπου του ΟΗΕ για την Άσον έχουμε ένα μικρό γραφείο περιφερειακό στη Μπανκόγκ που ασχολείται στη χώρα αυτή με τις 10 χώρες ΑΖΕΑΝ μαζί με τη γραμματεία ΑΖΕΑΝ και τους περιφερειακούς μηχανισμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΑΖΕΑΝ είχαμε γραφείο και στην Καμπότζη τα τελευταία 20 χρόνια ήταν από τα παλαιότερα γραφεία μας, στα επιτόπου στα πλαίσια της Συμφωνίας Ειρήνης του Παρισιού του 1983 και εξακολουθεί να ασχολείται με παροχή τεχνικής αρρωγής και υποστήριξη στον ειδικό εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη, μια εντολή που δημιουργήθηκε από την παλιά Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συνεχίστηκε στα πλαίσια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο Μιανμάρ λοιπόν μέχρι πρόσφατα ε, απ' έξω ασχολιόμασταν με τα ζητήματα αλλά με τις ταχείες μεταρρυθμίσεις ε, βελτιώσαμε και εμείς και αυξήσαμε την παρουσία μας στη χώρα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η οποία παρίσχε κάποια αρχική χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να εργαστούμε με τη νέα Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Μιανμάρ και πέρσι τον Νοέμβριο ο πρόεδρος Σάιν κάλεσε το γραφείο του είπα το εκπροσώπου να δημιουργήσει ένα γραφείο στη Μιανμάρ και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι γι' αυτό. Ξεκινήσαμε στις πραγματεύσεις με την κυβέρνηση σχετικά με τη συμφωνία με τη χώρα υποδοχής που θα είναι η βάση τέτοιου γραφείου. Δεν προχωρήσανε πολύ ακόμα οι διαπραγματεύσει, αλλά ελπίζουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία ίσως θα μπορέσει να προχωρήσει φέτος Εν τω μεταξύ, Κάνουμε τακτικές επισκέψεις στη Μιανμάρ από την Μπαγκόγκ και έχουμε τρία άτομα προσωπικό που βοηθούν τις ανθρωπιστικέ ε, υπηρεσίε στο έργο του. Και τέλος, μέχρι πρόσφατα, είμαστε ένα κομμάτι της αποστολή ενισχύσεως στο Ανατολικό Τιμόρ του ΟΗΕ. Ε, δεν εργαστήκαμε μετά την ανεξαρτησία. Ε, σιγά-σιγά μειώνεται η αποστολή στο Ανατολικό Τιμόρ που θα γίνει, είμαστε ακόμα εκεί και θα γίνει μέλος της ΑΖΕΑΝ πιθανότατα σύντομα. Έχουμε μερική αλλά συμμετοχή συμμετοχή σε εθνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο στις χώρες ΑΖΕΑΝ. Δεύτερον, θέλω να αναφερθώ στο τι γίνεται στους θεσμικούς μηχανισμούς και πλαίσια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή Άζεαν. Στις χώρες έχουμε τέσσερα θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις χώρες Άζεαν, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Μαλαισία. Όλα αυτά τα γραφεία, αυτές οι υπηρεσίες, έχουν καλό ιστορικό, έχουν πετύχει ε, ε, βαθμολόγηση επίπεδου α σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, συμμορφώνουμε τις αρχές των Παρισίων όσον αφορά τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρόμοιος θεσμός υπάρχει και στον Ανατολικό Τιμόρ, ένα είδος διαμεσολαβητή ε, είναι, αλλά έχει το ίδιο επίπεδο, την ίδια ισχύ όπως και μια υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το Μιανμάρ δημιούργησε μια επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωμάτων πέρσι ή τέλος του 2010 μάλλον ε, ε, λειτουργεί βάσει προεδρικού διατάγματος και διεξάγονται προσπάθειες, προσπαθεί να ε, θεσπιστεί νομοθεσία, μάλλον να υπάρξει σωστή νομοθετική πλαισίωση και συμμετέχουμε στην προσπάθεια ελπίζοντας ότι η σχετική νομοθεσία θα δώσει την κατάλληλη ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα στο φορέα, κάτι που απαιτείται σύμφωνα με τα επιτευθέντα σε κάποιες άλλες χώρες ΑΖΕΑΝ. Αυτά τα εθνικά θεσμικά όργανα είναι πολύ σημαντικά σε εθνικό επίπεδο, αλλά ξεκίνησαν να συνεργάζονται πολύ περισσότερο και σε περιφερειακό επίπεδο, παρέχουν υποστήριξη ο ένας φορέας τον άλλον, ασχολούνται με κοινά θέματα, ζητήματα κοινά που αφορούν τις χώρες ΑΖΕΑΝ. Δεύτερη σημαντική εξέλιξη αφορούσε την επέτειο των 40 ετών το 2009 των χωρών ΑΖΕΑΝ όπου το ΑΖΕΑΝ ε, υιοθέτησε νέα χάρτα ανανεωμένο όραμα του ΣΥΠΗΝ για τον οργανισμό αυτό και στη χάρτα συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά δέσμευση για συμμόρφωση με διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και ανθρωπιστικά πρότυπα και δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν τον πρώτο μηχανισμό, τον περιφερειακό για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ΑΖΕΑΝ. Θυμηθείτε ότι η περιοχή Ασίας και Ειρηνικού είναι μια περιοχή στον κόσμο που δεν έχει συγκεκριμένο περιφερειακό μηχανισμό για το ανθρωπίνο δικαίωμα, πλαίσιο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο με τους αντίστοιχους φορείς Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Είναι τεράστια περιοχή, ποικιλόμορφη, δύσκολο να επιτευχθεί, πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί το στόχος. Όμως ε, η Άζεν έδειξε ότι είναι εφικτό σε υποπεριφερειακό επίπεδο, σε μικρότερες συστάδες χωρών, να γίνει προσπάθεια για να δημιουργηθεί ο πρώτο περιφερειακό μηχανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα υπάρξει στην Ασία είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα, σημαντικότατο πείραμα. Συμμετείχαμε με θετικό τρόπο στην όλη προσπάθεια. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού που αποκαλείται διακυβερνητική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ΑΖΑΝ, ΆΙΤΣΑ, ήταν κάτι που προχώρησε πολύ γρήγορα, οι προδιαγραφές εσπίστηκαν πολύ γρήγορα, η εντολή που υθετήθηκε από τους ηγέτες και τώρα λειτουργεί και εφαρμόζεται από το 2010-2011. Αρχικό μοντέλο, αρχικό πρότυπο και εντολή του ΆΙΤΣΑ έχει κάποιους περιορισμούς, για να είμαστε ειλικρινείς. Νομίζω ότι τα βασικά κενά είναι τα εξή. Τα μέλη του ΑΙΑΤΣΑ είναι σε διακυβερνητικό επίπεδο. Οι εμπειρογνώμονε που διορίζονται είναι εκπρόσωποι κυβερνήσεων, δεν είναι ανεξάρτητοι επαείοντε, κάτι που βλέπουμε σε ευρωπαϊκού φορεί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι αφρικανικού φορεί ή α, ε, στο αμερικανικό, ε, της Αμερικανικής Υπήρου. Τα μέλη της ΑΕΤΣΑ είναι εκπρόσωποι κυβερνήσεων. Είναι διακυβερνητικό μηχανισμός. Ουχή περιφερειακός μηχανισμός, ανεξάρτητος. Και η εντολή είναι περισσότερο δίνει χαρακτήρα συμβουλευτικό στο φορέα. Δεν υπάρχει εντολή συγκεκριμένη για μέτρα προστασίας. Όπως άλλοι περιφερειακοί μηχανισμοί άρχισαν να δημιουργούνται και να ασχολούνται με διαφορετικά θέματα και ζητήματα σε επίπεδο χωρών όπως ανέφεραν από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τη Διεθνή Αμνηστία συνάδελφοι. Ασχολούνται με υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά η ΑΕΑΤΣΑ δεν κινείται σε επίπεδο προστασίας ατόμων, έχει γενικότερη, σφαιρικότερη προσέγγιση και το όμω, ελπίζουμε ότι η ΑΕΑΤΣΑ θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτή ήταν η εμπειρία μα από άλλε όπου κάθε περιφερειακός μηχανισμός, όπως και στην Ευρώπη, προόδευσε, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου και νομίζω ότι με τη σωστή ηγεσία, με τα σωστά μέλη, με τη σωστή διάδραση, με την κοινωνία των πολιτών, η ΆΙΤΣΑ μπορεί να ακολουθήσει παρόμοιο μονοπάτι και στο μέλλον. Η ΆΙΤΣΑ θα αναθεωρηθεί μετά την πρώτη τετραετία-πενταετία και αυτή θα είναι σημαντική στιγμή για προβληματισμό και ενδεχομένως για κάποιες αλλαγές και κάποιες βελτιώσεις ε, της ισχύουσας εντολής. Ταυτόχρονα η Άτσα δημιουργήθηκε ε, και μια επιτροπή για παιδιά και γυναίκες από τον Άζεν που έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το Άιτσα, αλλά κατά την αξιολόγησή μας ε, έχει μεγαλύτερο εύρος κινήσεων, ευρύτερη εντολή και μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας και μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο πείραμα. τουλάχιστον στη σφαίρα των δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών, ίσως να μπορέσει να δραματίσει ενεργότερο ρόλο από ότι η Άιτσα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικοί νέοι θεσμοί και νομίζω ότι είναι ένα σημείο σύνδεσης με το ευρωπαϊκό σύστημα, δηλαδή το σύστημα Άζια να συνδέεται κάπως με το ευρωπαϊκό, όσον αφορά τις δεσμεύσεις, ε, τυχόν υποστήριξη κλπ. Ένα από τα πρώτα βήματα του ΆΙΤΣΑ ήταν να αναπτύξει μια νέα διακήρυξη ΑΖΕΝ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χρειάστηκε και μια μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων μεταξύ ε, των ε, εκπροσώπων των κυβερνήσεων στην ΆΙΤΣΑ. Κατά την άποψή μας δεν υπήρξε επαρκή διαβούλευση και συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών τη περιφέρεια αυτή, τη περιοχή αυτή, να εκφράσουν την άποψή τους, ανησυχίες και προτεραιότητες και να ληφθούν υπόψη στο σχέδιο διακήρυξη. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο διακήρυξη που υθετήθηκε τελικά από τους ηγέτε πέρσι, εμπεριέχει σημαντικότατα στοιχεία, πολλά στοιχεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεσμεύσει. Υπάρχει ένα πληρέστατο φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται, σημαντικότατη δήλωση αρχών. Αν θέλετε η έλλειψη, το κενό που ενετόπισε ο ύπατος εκπρόσωπος ήταν το εξής, διτό πρόβλημα μάλλον. Πολλά από τα εμπεριεχόμενα δικαιώματα της διακήρυξης υπόκειται σε όρο ατυχή, πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με εθνικούς νόμους. Αυτό δίνει, πώς να το πω, δίνει ε, δημιουργεί ένα φραγμό όσον αφορά την πλήρη ερμηνεία των αρχών αυτών σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα για τα δικαιώματα. Και δεύτερον, ότι η διακήρυξη εμπεριέχει αρκετή έμφαση σε ευθύνε καθώ και τα δικαιώματα. Και ξανά και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητική ε, ερμηνεία σε, κάποιες, σε κάποια πλαίσια και περιπτώσεις. Αυτό που είναι σημαντικό ήταν ότι όταν θέτησαν ηγέτες Άζεν τη διακήρυξη στη διακήρυξη της ΠΝΟΜΠΕΝΧ δεσμεύτηκαν και είναι σημαντική δέσμευση ότι η διακήρυξη ΑΖΕΝ θα ερμηνευτεί και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις οπορέων της Διεθνής Συμβάσης και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των χωρών μελών. Οπότε αυτό είναι ένα μέτρο διαφύλαξης. Δηλαδή διακήρυξη ΑΖΕΝ, ναι μεν εμπεριέχει κάποιους περιορισμούς, αλλά πρέπει η ερμηνεία που δίδεται να ταιριάζει με τα διεθνή πλαίσια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δούμε η διακήρυξη ASEAN πώ θα χρησιμοποιηθεί, πώ θα προωθηθεί και πώ θα εφαρμοστεί στην πράξη από την ΆΙΤΣΑ. Σημαντικότατες εξελίξεις. Ένας από τους τομείς που έχει προτεραιότητα για την ΆΙΤΣΑ είναι η εταιρική ε, ευθύνη επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέποντας τη δουλειά που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εστιάστηκαν επί των, ευρωπαϊκ... των εθνικών θεσμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εθνικά σχέδια δράσης για τις επιχείρησεις τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέποντας όλα αυτά, αυτό θα μπορούσε ένα σημείο επαφής, διεπαφής μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων και του συστήματος ASEAN. Στρέφομαι τώρα προς κάποια βασικά θέματα που μπορούν να διατυπωθούν βλέποντας τις στάσεις και τη, τη δυναμική στις χώρες Άσεων. Ε, διάφορες συγκεκριμένες υποθέσεις αναφέρθηκαν τους συναδέλφους των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αρκετά από αυτά τα θέματα τελικά σχετίζονται με τη διαδικασία της δημοκρατικής αλλαγής ε, και παγίωσης της δημοκρατίας στην περιοχή. Ήταν μια περίοδος που διάρκεσε δύο, τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Πολύ σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν στις περισσότερες χώρες ΑΖΕΑΝ, το Βιετνάμ και το Λάος εξακολουθούν να έχουν μονοκομματική δομή, αλλά στις περισσότερες από τις άλλε χώρε είδαμε μια επέκταση, εξάπλωση των ε, δημοκρατικών θεσμών, του δημοκρατικού χώρου, ανάπτυξη νέων δημοκρατικών θεσμών. Το Μιανμάρ είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Ε, το Μιανμάρ περνάει μια πάρα πολύ σημαντική πολιτική μετάβαση και αλλαγή, αλλά και ακόμα πιο εδρεωμένε δημοκρατίες ακόμα και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει μια δυναμική που δημιουργεί προβλήματα οι δικαιώματα. Στην Ταϊλάνδη, ε, οι πτυτικές εξελίξεις, ε, πολύ γρήγορες αλλαγές, πόλωση πολιτική τελευταία περίοδο που δυστυχώς οδήγησε σε πολιτική βία το 2010 η Ταϊλάνδη ε, δημιούργησε με επιτροπή συμφιλίωσης και εξυχνίασης. Πολύ σημαντικό, παρά τους περιορισμούς, συνέταξε καλή έκθεση που απέδωσε ευθύνες ε, και οδήγησε και πρότεινε σημαντικέ θεσμικέ μεταρρυθμίσει. Κάτι που ενθαρρύνω μετά μάλλον όσον αφορά τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί σε αυτή την έκθεση. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον τη ε, Ταϊλάνδη. Και στη Μαλαισία λοιπόν, όπου το πολιτικό περιβάλλον επισκιάστηκε επί μακρόν για διάφορους, από διαφόρους νόμους για την ασφάλεια, περιορισμό για δημοσιεύσεις. Ε, πριν από ένα-δύο χρόνια ένα, ένα κίνημα για ελεύθερες εκλογές ή ένα περιβάλλον για ελεύθερες εκλογές ε, καταπιέστηκε, αντιμετώπισε κυρώσει. Είδαμε αρκετά σημαντικέ εξελίξει όσον αφορά την κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση ανέξε νέου χώρου, κατήργησε κάποιου από του ε, νόμου περί ασφαλείας, Παρόλο βέβαια που εισήγαγε κάποιε περιοριστικέ διατάξει μέσω θέσπιση νέα νομοθεσία, παρόλα αυτά όμω είναι σημαντικέ οι αλλαγέ που σημειώθηκαν και πρόσφατα είδαμε να έδωθεί και άδεια για διαδηλώσει αντιπολίτευση και να δημιουργηθεί νέο χώρο, νέα δυνατότητα κίνηση. Στην Ινδονησία επίση, όπου επί μία δεκαετία και παραπάνω από δεκαετία έγιναν σημαντικές αλλαγέ, παγιώθηκε η δημοκρατία, οδηγείται προς άλλο κύκλο προεδρικών εκλογών θα λάβουν χώρα του χρόνου. Παρόλα αυτά, εντάσει, τάσει αφορούν περισσότερο τον τομέα τη ευτική ανοχή και το παρατήρησε η ΥΠΑΤΗ Επίτροπος όταν επισκέφθηκε τον Νοέμβριο πέρσι ε, την Ινδονησία. Υπάρχει βιο, υπάρχουν βιοπραγίες κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, Σιαΐτες, Χριστιανοί, Αμάντι. Ε, υπάρχουν ε, περιορισμοί που πλευράλλονται από το κράτος στη μειονότητα Αμάντι και αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις για τις λαϊκές παραδόσεις της χώρας ε, και το θέμα της σκεπτικής ανοχής που θέλουν να επικρατεί στη χώρα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Η ελευθερία της έκφρασης ε, είναι προβληματική. Αναφύεται, το είπε και η Διεθνής Αμνηστία και η Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, καταδικάστηκαν δημοσιογράφοι και bloggers στο Βιετνάμ ή ε, χρησιμοποιήθηκε ο νόμος κατά επικριτών της κυβερνήσης του Ταϊλάνδη, χρήση νόμων περί συκοφαντίας στην ε, Καμπότζη κατά ακτιβιστών και μελών της αντιπολίτευσης που αναφέρθηκαν τους συναδέλφους και ακόμα χειρότερος ακραίες περιστάσεις έχαμε φόνους και εξαφανίσεις ε, προσπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ακτιβιστών του περιβάλλοντος ή για κοινωνικές αλλαγές σε διάφορες χώρες. Πιο πρόσφατα είδαμε την υπόθεση στο Λάος που προβλήθηκε πάρα πολύ του κύριου Σολβατσον Πον. Αυτά επίσης ε, συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με κάποιες από τις ε, υποφόσκουσες συγκρούσεις στην περιοχή ή στις ζώνες συγκρούσεων που εξακολουθούν υπάρχουν συγκρούσεις, βιοπραγίες στη Μιανμάρ, στο κράτος Ρακάν, Καντσίν και στην Πάπα Ινδονησία, Νότια Ταϊλάνδη και τώρα στις Φιλιππίνες ε, ε, ευτυχώς υπήρξε νέα ειρηνευτική συμφωνία όπου παρόλα αυτά όμως συνεχίζονται οι βιοπραγίες. Ανέφερα και άλλα δύο θέματα. Αναφέρω σύντομα δύο άλλα θέματα, μια και πιέζει ο χρόνο, που ίσω δεν έτυχαν τη προσοχή μα. Η μετανάστευση ένα από αυτά. Πολύ περίπλοκο, σύνθετο θέμα για αυτή την υποπεριφέρεια. Αυτέ οι χώρε είναι και πηγέ ταυτόχρονα εργαζομένων εξωτερικά, αλλά είναι και χώρες υποδοχής εσωτερικά και υπάρχει και μεγάλη ροή, μεταναστευτική ροή σε σχέση με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Είναι επίσης μια σημαντική διακομιστική, διαμετακομιστική περιοχή διόδου και για πρόσφυγες και για ετούντες άσυλο. Και σημαντικές κινήσεις σημειώνονται αυτή τη στιγμή προς την Ταϊλάνδη και στη συνέχεια προς την Μαλαισία. Σε κάποιες περιπτώσεις επίσης ετούντες άσυλο περνούν με λαθρεμπόρους μέσα από διάβλους ε, και κινούνται σε χώρες τελικά, τελικού προορισμού όπως η Αυστραλία. Όλο και περισσότερη συζήτηση γίνεται για ένα θεσμικό περιφερειακό πλαίσιο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων πλέον. Και ένα από τα κενά που υφίστανται είναι, αν θέλετε, η έλλειψη επικύρωσης ε, της σύμβασης για τους πρόσφυγες ε, σε πολλές από τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας ε, για αυτού του είδους τους ανθρώπους που διακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια σημαντική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εμπλακεί υπό τους όρους της δικής της πείρας σε σχέση με τις περιφερειακές αυτές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των θεμάτων ασύλου. Και η θανατική ποινή εν τέλει, και το αναφέρανε αυτό πιο πριν, είναι ένας ενδιαφέρον τομέας αυτός, όπου δεν σημειώνεται πρόοδος μέσα στο πλαίσιο των χωρών ΑΣΕΑΝ είναι χώρες τόπου, η πρώτη γραμμή για την θανατική ποινή. Έχουμε κάποιες από τις πιο ισχυρές ε, χώρες για την κατάργηση Φιλιππίνες, ε, Καμπότζη και κάποιες από τις πιο ισχυρές διατήρησης της θανατικής ποινής όπως η Σιγκαπούρη για παράδειγμα. Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν κάποιες ενδιάμεσες χώρες όμως στο ενδιάμεσο πλαίσιο που διατηρούν τη θανατική ποινή κάποιες χρονικές περιόδους ε, και υπάρχουν και μορατόρια μακρότερης διάρκειας όπως στην ε, Ταϊλάνδη για παράδειγμα αλλά και για την Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις που σημειώνονται να αποκλίνουν από την ε, επιβολή, υποχρεωτική επιβολή της θανατικής ποινή και να ξεκινήσουν κάποιες συζητήσεις σε σχέση με το ζήτημα της θανατικής ποινή μικρά αλλά σημαντικά βήματα παρόλα αυτά προς την σωστή κατεύθυνση της, ε, τουλάχιστον του περιορισμού τουλάχιστον ε, της εμβέλειας ε, του φάσματος επιβολής της θανατικής ποινής και μιας απόκλησης από αυτή την κατάσταση προς τους στόχους που προασπίζεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Αυτή είναι η δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. you all. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές γιατί μας παρουσιάσατε πολλά θέματα και μας κάνατε και πλήρη ανάλυση ώστε τώρα έχουμε όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που είπατε για την Επιτροπή ΑΣΕΑΝ για, την, για τις γυναίκες και τα παιδιά. Αυτή η Επιτροπή βρίσκεται στις Βρυξέλλες και ζήτησαν να παρευρεθούν ε, ζητήσαμε εμείς να παρευρεθούν, αλλά δεν δέχτηκαν την πρόσκλησή μας, γιατί θεώρησαν ότι δεν ε, είναι τμήμα ε, της δραστηριότητάς τους να έρθουν σε μια επιτροπή σαν τη δική μας. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι περιορισμοί και στο ποιους μπορούμε να έχουμε κοντά μας για να συζητήσουμε. Θα θέλαμε να είναι παρόντες, αλλά δεν ε, κατέστη δυνατόν. Όσον αφορά ε, τους θεσμικούς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εσείς αναφέρετε ε, κάποιους θεσμούς που αναπτύσσονται ή που ήδη υπάρχουν στην Ασία. Στην Επιτροπή μας συχνά αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα και σήμερα το απόγευμα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με από χώρες της Ανατολικής ε, συμμαχία τη Ανατολικής Ευρώπης και βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, ε, προδιαγραφές και διαφορετικά standards ακόμη και σε χώρες της Ευρώπης. Περιγράψατε ως καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου να ασχοληθούμε με το θέμα των προσφύγων και των μεταναστών στην Ασία. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Νομίζω ότι δεν έχουμε απολύτως τη δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν έχουμε ε, τη δυνατότητα ε, επικύρωσης θεμάτων που αφορούν τους πρόσφυγες και τις μειονότητες και τις οικογένειές τους. Επομένως, έχουμε και εμείς πράγματα που ακόμη μπορούν να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, πολλά κρατημέλη που δεν συμφωνούν με την επικύρωση, παρότι συμφωνούν με πολλές από τις συστάσεις. Τώρα, ο κύριος Ανιέρη Σαμπατούκη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, υπεύθυνο της ε, Διεύθυνσης ΑΣΕΑΝ. και οι δύο εκπρόσωποι από την Διεθνή Αμνηστία και από την ε, Διεθνή Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκαν ε, σε αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να ακούσουμε και εσάς, να μας πείτε πώς το βλέπετε εσείς από τη δική σας οπτική γωνία και τι κάνετε εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς ερχόμουν εδώ σε σχέση με την εκπροσώπηση του Γραφείου για την Νοτιοανατολική Ασία και καθώς ε, αναμενόταν παρέμβαση σε σχέση με τα θέματα ξεχωριστά αυτών των χωρών από το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτό δείχνει την θέση που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη σχέση μας ε, με τις χώρες ε, των, της Νοτιοανατολικής Ασίας που έχει μεγάλη σημασία το θέμα Ουσιαστικά θεμελιώνουμε την ημερήσια διάταξή μας ε, στο έργο για τα δικαιώματα υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου και σε συζητήσεις και επαφές με την κοινωνία των πολιτών και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο και φυσικά ε, έχουν ε, μεγάλη σπουδαιότητα αυτοί οι εταίροι μας σε αυτή τη διαδικασία συνολικά. Όπως είπα, τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι ένα από τα πιο σημαντικά και εμβαθυμένα πεδία στις σχέσεις μας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας καλύπτουμε τις δραστηριότητες μας αυτές μέσω πολυσχηδών μέσων και εργαλείων. Από τότε που ανέλαβα από την 1η Οκτωβρίου 2012 αυτά τα καθήκοντα πέρυσι, εντυπωσιάστηκα πολύ από το έργο που επιτελείται σε αυτό το πεδίο, που θεωρώ ότι είναι αναλογικά ακόμα μεγαλύτερο από αυτό το οποίο επιτελείται σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου σύμφωνα με την πείρα μου. Έχουμε έναν αριθμό ε, τυπικών και επίσημων διαλόγων, άτυπων και επισήμων ταυτόχρονα. Με έξι χώρες έχουμε αυτό το διάλογο που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Έχουμε ένα που διεξήχθη πριν από λίγες ημέρες κιόλα ε, σε σχέση με το Λάος έχουμε σημαντικές διατάξεις και προδιαγραφές για τα δικαιώματα του ανθρώπου στις διάφορες PCAs, δηλαδή τις ε, ε, Partnerships and Cooperation Agreements, συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, και συνεργασίας με τις περισσότερες από αυτές τι χώρε της Νοτιοανατολικής Ασίας. Κατά τις διμερείς μας συναντήσεις γνωρίζετε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα πάγιο σημείο ανταλλαγή απόψεων και αναφέρθηκε και το θέμα σε σχέση με την Καμπότζη όσον αφορά τα θέματα γεωκτησίας για παράδειγμα στην Καμπόζη όταν ο πρόεδρο του Συμβουλίου, Χέρμαν Φαν Ρόμπα, πήγε στην Καμπότζη πέρσι τον Νοέμβριο, το έθιξε αυτό το θέμα, το ανέφερε σε σχέση με του ομολόγου του εταίρου τη Καμπότζη. Και ένα σημαντικό μέρο τη συζήτηση ε, εκτελήθηκε γύρω από, γύρω από αυτόν τον άξονα. Γνωρίζουμε ότι ο Επίτροπο Ντεχούχτ, όταν θα πάει ε, τον Μάρτιο για την οικονομική διάσκεψη κορυφή ε, ΑΣΕΑΝ και σε σχέση με αυτά τα θέματα και πάλι θα συζητήσει και θα θίξει αυτό το συγκεκριμένο, αυτά τα τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και έχουμε και συγκεκριμένα διαβήματα που βρίσκονται υπό εξέλιξη. Οποτεδήποτε πάντα θεωρούμε ότι είναι εύθετο να γίνει αυτό. Είχαμε μια τέτοια επαφή και εξέλιξη με το Λάος σε σχέση με το ζήτημα της αντιμετώπισης ε, του, των δικαιωμάτων του α, υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σομπα, σου, που αναφέρθηκε προηγούμενα και από εσάς που είναι ένα θέμα που μας απασχολεί τα μάλα Επίσης, σε σχέση με τους όρους ε, κάποιων δηλώσεων που προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε πολυσχηδή προγράμματα και σχέδια μέσω της κοινωνίας των πολιτών και μέσω των, της συμμετοχής και σε σχέση με κυβερνήσεις, κυβερνητικούς εταίρους που είναι εταίροι μας σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Προηγούμενα αναφέρατε επίσης και μάλιστα μας ικανοποιεί αυτό το ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία μπορούμε να καλωσορίσουμε την ε, προσπάθεια που γίνεται για την προστασία των δικαιωμάτων γυναικών και παιδιών. Αυτή η αντιπροσωπεία βρίσκεται εδώ στις Βρυξέλλες και είχαν και μια συνάντηση με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη από χθες και επισκέπτονται και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα καθώς επίσης και ε, βέλγικούς θεσμούς. Δεν έχω όλες αυτές τις λεπτομέρειες γιατί μόλις ξεκίνησε αυτή η επίσκεψη από πλευρά τους. Αλλά από ό,τι γνωρίζω είναι πραγματικά σε βάθος και ε, έντονες συζητήσεις, ζωντανές συζητήσεις. Αυτό αφορά και την ε, Επιτροπή σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου που προσήλθε στις Βρυξέλλες ήδη το 2011. Όλα αυτά συνολικά τι θέλουν να κάνουν. Να δώσουν μια προοπτική να ενταχθούν στο πλαίσιο, σωστό πλαίσιο αυτές οι σχέσεις μας που είναι σύνθετες και περίπλοκες, ε, πολυσχηδείς και πυκνές με πολλά και διαφορετικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να καλλιεργήσουμε αυτές τις σχέσεις. Ε, σε σχέση με την Καμπόζη για παράδειγμα, να αναφέρω εδώ το ότι πράγματι καμιά φορά πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν κάνουμε λόγο για μέσα και εργαλεία, αν κάποιες από τις λύσεις που προτείνονται θα μπορούσαν εν δυνάμει μήπως να αντιστρέφονται και να αντιβαίνουν τις προσπάθειες υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Οι ε, προτιμήσεις, εμπορικές προτιμήσεις ε, για την Καμπόζη βοήθησαν σε πολύ μεγάλο, σε τεράστιο βαθμό τη χώρα να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τις ε, προδιαγραφές για την ευημερία της αυτής της χώρας. Διπλασιάστηκε το ανακεφαλήν εισόδημα και διεξάγοντας αυτές τις συζητήσεις πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κάποια από αυτά τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται όταν καταργούνται, όταν παγώνουν, ίσως μπορούν να συνεπάγονται και το πάγωμα ή την επιδίνωση και υποβάθμιση των κεκτημένων και έχουμε λοιπόν διατάξεις ώστε να μπορούμε να εντάσσουμε όταν έχουμε αυτές τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας στην ρήτρα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το πάγωμα αυτής της ρήτρας αν κάποιες χώρες δεν συμμορφώνονται αλλά αυτό είναι το ίστατο μέσο το ίστατο στο οποίο μπορούμε να προσφύγουμε. Και σε σχέση με την αναφορά που έγινε προηγούμενα για την ε, σημασία, τη σπουδαιότητα τη ε, ε, διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου του Νοεμβρίου 2012, γνωρίζουμε ότι αυτό δημιούργησε ευρύτερε συζητήσει μέσα στο πλαίσιο τη διεθνού κοινότητα ω επίμαχο θέμα και με του εταίρου τη Νότια Νότιας Ασίας. Υπάρχουν ανησυχίες που εκφράστηκαν για τον κίνδυνο της πρόκλησης της οικουμενικότητας και εμεί εξετάσαμε εξετάσαμε αυτή τη διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου πάρα πολύ προσεκτικά και είχαμε σε βάθο συζητήσει εσωτερικά. Αποφασίσαμε να δούμε και να πούμε ότι το ποτήρι είναι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Να δείξουμε δηλαδή κάποια αισιοδοξία. Θα ήταν ε, εκτό ε, κάθε φαντασία το ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί όπως βλέπαμε τα πράγματα πριν από λίγα χρόνια, μια τέτοια διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου από αυτές τις χώρες. Είναι λοιπόν μια καλή θετική βάση επί της οποίας μπορούμε να εργαστούμε και να προσφέρουμε στους εταίρους μας της Νότιας Ασίας, Νοτιοανατολικής Ασίας τις ε, δυνατότητες να εφαρμοστούν όλα αυτά στο δυνατό του εφικτού κατά το μέγιστο βαθμό, ώστε η οικουμενικότητα όλων των πτυχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου να είναι σεβαστή πανταχώθεν και σε όλες τις πλευρές της. Έχουμε λοιπόν μια θετική βάση εργασίας και συνεργασίας, ώστε να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε για τα δικαιώματα του ανθρώπου στο περιφερειακό πλαίσιο, που είναι και αυτό σημαντικό για τη σχέση μας. Θέλουμε να αυξήσουμε, σημαντικά κιόλα να αυξήσουμε την δέσμευσή μας υπέρ αυτών των, της ευδοκίμησης αυτών των στόχων με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας Φυσικά αναφέρατε κάποιες ατομικές περιπτώσεις επιμέρους χωρών και ατομικών περιπτώσεων. Δεν θα τις απαριθμίσω όλες αυτές. Είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε και να τοποθετηθούμε διμερώς σε οποιαδήποτε παρέμβασή σας γιατί διαφορετικά θα αναλώναμε υπερβολικά πολύ χρόνο. Ιδιαίτερα ε, ε, είχαμε εμπλακεί κατά το τελευταίο διάστημα για την κατάσταση ε, του υπέρμαχου Σομπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ήδη το Δεκέμβριο ζητήσαμε να αναλυθούν δοθούν ε, διαβήματα και να γίνει κάτι γι' αυτόν. Είχαμε επαφές με κυβερνητικού εκπροσώπους και μάλιστα και σε καθημερινή βάση προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να συζητήσουμε και να δούμε με ποιον βέλτιστο τρόπο θα μπορούσαμε να συνδράμουμε, να παράσχουμε την ε, ε, συνδρομή μας και να εμπλακούμε ώστε να έχουμε μια το δυνατόν θετικότερη απάντηση. Δυστυχώ. δεν έχουμε υπερβολικά πολλά καλά μαντάθα να σας αναφέρουμε, αλλά παρόλα αυτά υπήρξε μια, ένας ρόλο ρόλος από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθήσαμε να διαδραματίσουμε ως ΕΕ στα διαβήματα τα οποία αναλύθηκαν έγιναν όλα αυτά όχι μόνο εξ ονόματος Ε, ΕΕ αλλά και εξ ονόματος των διεθνών εταίρων όπως της Αυστραλίας, των ΙΠΑ και της Σιγκαπούρης που είναι η πρώτη ε, χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας ε, που προσέθεσε τις προσπάθειές της στο πλευρό των δικών μας σε αυτά τα διαβήματα. Προσπαθούμε στο βαθμό του εφικτού να συνεργαστούμε με τους ε, εταίρους μας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας να δούμε τι μπορεί να επιτευχθεί. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ένας αριθμός κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν προχωρήσει και έχουν στο Βιεντιάνε, στο λαό για να συζητηθεί αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση αυτά, αυτό το θέμα είναι καλά μαντάτα αυτό ιδιαίτερα σε σύγκριση με το τι συνέβαινε πριν από κάποια χρόνια στο παρελθόν φυσικά πολλά άλλα θέματα αναφέρθηκαν και είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε και να τοποθετηθούμε στις επαφές μας διμερό. Ευχαριστώ Thank you. Ευχαριστώ Τα μέλη μπορούν να πάρουν το λόγο αν επιθυμούν Δεν βλέπω να θέλει κάποιος. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις, απευθυνόμενοι προς εσάς επίσης. Ο κ. Μαγκόουαν είχε προτείνει στο μέλλον να εστιαστούμε περισσότερο ε, στην περιοχή, ε, περισσότερο να εστιαστούμε στο θέμα των επιχειρήσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύετε κι εσείς το ίδιο? Έχε, θεωρείτε ότι κι εσείς ότι αυτό είναι ένα δεχόμενο. Και δεύτερον, Ήταν πολύ καλή χειρονομία από την πλευρά σας. Εκονίσατε συνάντηση όταν έγινε ο διάλογος Βιετνάμ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρχει δυνατότητα μέλη της Επιτροπής ΔΡΟΑ να έχουν άμεση ανταλλαγή απόψεων με, του, με την αντιπροσωπεία του Βιετνάμ. Ήταν πολύ καλή εμπειρία. Μάθαμε πράγματα. Έμαθα πράγματα. Όμως έχω κάπως διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχω ανοιχτή ανταλλαγή επιστολών με τον κύριο Ντεκούχτ. Ε, ξέρω ότι δεν υποστηρίζω απόλυτα την προσέγγιση του, κυρίως όσον αφορά την εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ που συζητείται. Αφορά περισσότερο να μην μένουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτός του πλαισίου των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Βιετνάμ, αλλά γενικά. Υπάρχουν εμπειρικές αποδείξεις που λένε ότι όταν έχει αύξηση του εμπορίου και καλύτερες οικονομικές συνθήκες, θεωρείται ότι αυτομάτως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα βελτιώνονται. Αυτό θεωρείται. Βεβαίως, εγώ δεν είμαι κατά του εμπορίου. Το δικαίωμα για τη στέγαση, για την τροφή είναι σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα και μπορούν να βελτιωθούν, αλλά πρέπει να δούμε και αν αλλάζει η κοινωνία. Υπάρχουν διάφορες ομάδες στην κοινωνία που μπορεί να χάνουν από την όλη διαδικασία. Ε, ίσως να παραβιάζονται άλλα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην κοινότητά μας Ευρωπαϊκής Ενώσης χρειάζεται περισσότερη συζήτηση. Το ίδιο ισχύει και στο Κοινοβούλιο. Κύριε Τσίπ, νομίζω ότι η γνωμοδότησή σας για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή η εταιρική κοινωνική ευθύνη ήταν το θέμα. Ε, ετοιμάσαμε πολύ καλή γνωμοδότηση, τη στείλαμε στις δύο επιτροπές μας και οι αντιδράσεις ήταν αντίθετες των δύο επιτροπών, αντίθετες μεταξύ τους. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι κάτι μόνο για κήρυγμα κυριακάτικο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να εφαρμόζεται, να λαμβάνεται υπόψη για να βελτιώνεται και η διαμόρφωση της πολιτικής. Το πιστεύετε κι εσείς αυτό. Αυτά που έλεγε την ανταλλαγή επιστολών με τον κύριο Ντεκούχτ, ε, εντάξει, αυτό ήταν απλώ για ενημέρωσή σα, δεν ήταν ερώτηση. Θα μπορούσατε όμω να απαντήσετε στην προσοχή που πρέπει να δοθεί στην περιοχή αυτή, στις επιχειρήσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Είναι μια όλο και περισσότερο σημαντικότερη πτυχή αυτή και πράγματι μέσω του είδου εμπλοκή ε, που έχουμε μέσω του, των PCA, των Συμφωνιών εταιρική Σχέση και Συνεργασία, είναι ένα μεγάλο κουτί κυβότιο όπου όλου του είδους, ό, όλων των ειδών οι πολιτικές εντάσσονται σε αυτό και είναι μια ευκαιρία να δράσουμε και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την εγκάρσια, την οριζόντια πολιτική και διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών πτυχών αυτών των πολιτικών. Τώρα όσον αφορά την εταιρική ευθύνη. Είχαμε ένα σεμινάριο πρόσφατα στην Ταϊλάνδη σχετικά και επίσης εξετάζουμε υποστηρικτική δράση στη Μιανμάρ για παράδειγμα σχετικά με αυτό το πλαίσιο. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Είναι πολύ σοβαρά, είναι πάρα πολύ σημαντικά υπό την πτυχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και σημαντικά όλα αυτά για την πτυχή των εμπορικών σχέσεων για το εμπόριο έχουν επιπτώσεις όσον αφορά στο πω έτσι ένα ισοδίκαιο πλαίσιο, πεδίο δραστηριοποίησης. Προφανώς έχει πολύ σημαντικά στοιχεία υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Λαμβάνεται υπόψη να φωτέρωθεν αυτό και από τις δύο πλευρές το εξετάζουμε. Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα, να μπορέσουν περισσότερα να επιτευχθούν. Δεν έχω όλο τον κατάλογο των σχεδίων και ε, δράσεων των προγραμμάτων μας, αλλά πρόσφατα έχουμε πολλά κάνει και συνεχίσουμε αυτή την κατεύθυνση προς το μέλλον. Αν ενδιαφέρεστε μπορώ να σας διαθέσω περισσότερο εκτεταμένα και λεπτομερή στοιχεία για αυτή την παρουσίαση αυτού του θέματος. Πώς εντάσσουμε αυτές τις σημαντικές πτυχές στις συζητήσεις μας. Um, yeah, we have time for a change. That... Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο για ανταλλαγή απόψεων και ο πρέσβης της Μαλαισίας έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Πρέσβη, νομίζω ότι έχετε ήδη ενημερωθεί ότι στην Επιτροπή μας ο κανονισμός λέγει ότι στους πρέσβεις δίνουμε τρία λεπτά χρόνο ομιλίας. Έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο σήμερα, αλλά θα σας παρακαλούσα να μην ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μας δίνει τη δυνατότητα και σε μένα και στους άλλους συναδέλφους να παρευρεθούμε σε αυτή τη συνεδρίαση. Και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Όντως έχω ενημερωθεί ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο ομιλίας. Μου το είχαν πει και πριν από τη συνεδρίαση. Παρότι πιστεύω ότι το θέμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Και δεν θα επαναλάβω τα θέματα τα οποία ήδη αναφέρθηκαν από τους εμπειρογνώμονες. Χαίρομαι που άκουσα τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων και των εκπροσώπων της Διεθνούς Αμνηστίας που αναγνώρισαν ότι υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις στη Μαλαισία και στην γενικότερη περιοχή ε, των χωρών ΑΣΕΑΝ όσον αφορά τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, δεν θέλω να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για τα σχόλια που έκανε η Διεθνής Αμνηστία συγκεκριμένα για τη θανατική ποινή και για την ελευθερία έκφρασης. Αρκεί νομίζω να πω ότι η κυβέρνηση της Μαλαισίας πιστεύει στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Και όπως είπε και ο επικεφαλής του τμήματος ε, Ασίας Ειρηνικού του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών ε, στη Γενέβη, προσπαθούμε να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις. Και είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε με τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να βελτιώσουμε την κατάσταση στη χώρα μας. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, όπως είπαν κάποιοι εμπειρογνώμονες, και εμείς είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Και η σημερινή συζήτηση είναι πολύ χρήσιμη. Ελπίζω να συνεχίσουμε μια τέτοιου είδου συζήτηση εδώ ή σε κάποια άλλα βήματα και θα είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τα θέματα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν. Να ξέρετε ότι η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή και αν υπάρχουν θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε, εγώ ευχαρίστως θα τα συζητήσω μαζί σας. Νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα προωθήσουμε την καλύτερη κατανόηση μεταξύ μας. και το σωστό είναι να χρησιμοποιήσουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς αν υπάρχουν οποιασδήποτε διαμαρτυρίες ή διαφωνίες νομίζω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε και αυτό είναι ο κατάλληλος διάβλος για τις συζητήσεις. Και μιας και έχω το λόγο θα ήθελα να πω κάτι γιατί αναφέρθηκε από κάποιον εμπειρογνώμονα η διακήρυξη των δικαιωμάτων για τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Είμαστε ακόμη ε, στο στάδιο που διδασκόμεθα και σίγουρα υπάρχει πεδίο βελτίωσης και από καιρούς καιρών πρέπει να γίνεται κάποια επανεξέταση και αναθεώρηση. Όπως είπατε και εσείς, βρίσκονται ε, στις Βρυξέλλες εκπρόσωποι της ACWC και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που δίνετε να γίνει αυτή η επίσκεψη. Ο σκοπός είναι να διδασκόμεθα από εσά, να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων και να προσπαθούμε να μαθαίνουμε τις βέλτιστες πρακτικές από εσά. Ξέρω ότι δεν έχω περισσότερο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη. Υπάρχει κάποιος άλλος. Ο κύριος Τσίπ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαγκόβερν, διότι στην παρουσίαση που έκανε σχολίασε εν γέννη τα διάφορα ζητήματα και αναφέρθηκε σε κάποιες πτυχές. Αναφέρθηκε στην κοινωνική εταιρική ευθύνη. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια πλατφόρμα, μια βάση όπου ο ΙΕ όταν καθόρισε κατευθυντήριες γραμμές ε, συζήτησε σφαιρικά το θέμα θεωρητικά. Όχι μόνο για μερικές χώρες. Είναι κάτι που αφορά όλες τις χώρες μέλη του ΟΗΕ. Το ζήτημα αυτό της εταιρική ευθύνης, κοινωνικής ευθύνης. Συνεχίζοντας λοιπόν από αυτό, πρέπει να πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενστερνίζονται αυτή την προσέγγιση, αλλά και στις σχέσεις μας με εταίρους σε διάφορα πλαίσια συνεργασίας, αυτό αποτελεί θέμα συζητήσεων. Χάρη στην προαναφερθή γενική προσέγγιση. Εγώ βλέπω δύο συναφή ζητήματα που είναι σημαντικά. από τη μία πλευρά έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. από την άλλη πλευρά έχουμε το θέμα του εμπορίου, των επιχειρήσεων, της οικονομικής δραστηριότητας, εν τη ευρία ενία του όρου. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση. Μια σχέση με την πρακτική εφαρμογή όλων αυτών, με την πρακτική διάσταση. Πρέπει να προωθούμε δραστηριότητες τέτοιες, όπου επιχειρηματική κοινότητα, επιχειρηματικός κόσμος, να βοηθά τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων για να παρατηρείτε πώς η τήρηση των κανόνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και πώς μπορούν να βελτιωθούν οι σχετικές προδιαγραφές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και απ' την άλλη πώς ίσως μπορεί να δημιουργούνται εμπόδια για την, ε, όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι εμπορικές σχέσεις μπορεί να επηρεάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια εταιρεία που χρησιμοποιεί τα παιδιά σαν σκλάβους για να παράγουν προϊόντα ή κάποια εταιρεία που πληρώνει με πολύ χαμηλές αμοιβέ τους εργαζομένους. Είναι ένα άλλο παράδειγμα. Αυτέ οι επιχειρήσει παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα, μπορεί να ανταγωνίζονται άλλε εταιρείε που προσπαθούν να συμμορφώνονται με τι υψηλέ προδιαγραφέ που επιβάλλει ο Διεθνή Οργανισμό Εργασία. Θέλουμε να είναι ο ανταγωνισμό θεμητό και δίκαιο. Αλλά πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αυτό το πλαίσιο και η ανθρώπινη διάσταση. Έχουμε κατευθυντήριες γραμμές στο ΙΕ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Απ' την άλλη έχουμε το Εθνές Γραφείο Εργασίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΣΑ, που όλοι προσπαθούν να κινηθούν στο σωστό πλαίσιο, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνη των επιχειρήσεων. Υπάρχουν λοιπόν σημεία επαφής μεταξύ των διαφόρων φορέων. Οι αρχές αυτές λοιπόν και οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούν να συζητώνται σε διάφορες διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα. Πώς μπορεί να υποστηριχθεί η όλη προσέγγιση. Αναφερθήκατε σε, διάφορους, ε, σε διάφορα θεσμικά όργανα διεθνή που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπου υπάρχουν αυτοί οι φορείς. Και όπου υπάρχουν τέτοιοι περιφερειακοί θεσμοί πρέπει να συμμορφώνονται με διεθνείς προδιαγραφές αυτοί οι φορεί μπορεί να βοηθήσουν στο να εφαρμόζονται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο οι διεθνεί προδιαγραφέ και ε, οι διάφοροι κανόνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, για τη μετανάστευση. Επανειλημμένα κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα. Είναι κάτι που αφορά και την Ευρώπη. Οι περισσότεροι μετανάστε πάνε συνήθω σε πλούσιε χώρες της Μέση Ανατολής Συχνά λοιπόν πάνε σε χώρες όπου ίσως δεν μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις σκεφτικές τους πεπιθήσεις. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή. Κάποιες χώρες επιτρέπουν, επιτρέπουν τη θρησκευτική λατρεία ελεύθερα. Άλλες χώρες έχουν συνταγματικό πλαίσιο που εμποδίζει κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Πιστεύω ότι η δραστηριότητα του ΟΗΕ και η δική σας δραστηριότητα δημιουργεί τη δυνατότητα να, να υπάρξουν πιέσεις για αλλαγές με την πάροδο των ετών. Είναι σημαντικό για κάποιον που μεταναστεύει όχι μόνο να μεταναστεύσει και να βρει ε, δουλειά και να μπορεί να δουλεύει ελεύθερα, αλλά όταν δουλεύει, να δουλεύει σύμφωνα με τι διεθνεί προδιαγραφέ για την απασχόληση. Να μπορεί ο άνθρωπο αυτό να ζει αξιοπρεπώ στη χώρα μετανάστευση. Να μπορεί ο μετανάστη να απολαμβάνει πλήρω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του. Να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα σαν άνθρωπο. Λοιπόν, το τελευταίο που είπατε, λέει Πρόεδρο, ότι θα πρέπει να εστιαστούμε και επί των δικαιωμάτων των μεταναστών και των οικογενειών του, ανεξάρτητα από το που βρίσκονται. Έχουμε πάντα στην Επιτροπή μας ε, το θέμα αυτό προς συζήτηση. Μπορούμε να το θέτουμε αυτό και όταν γίνεται ανταλλαγή απόψεων με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και με άλλες περιοχές. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να συγκεραστούν όλες οι πτυχές και όλοι οι συνομιλητές. Πολύ συχνά γίνονται προσπάθειες με μονομένες χώρες. Έγινε μια ακρόαση για το Κατάρ την προηγούμενη φορά στην Επιτροπή. Χρειάζεται συστηματικότερη προσέγγιση, πιστεύω. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου άποψη. Αυτά έχω μάθει. Ε, θα ήθελα να δώσω στους εμπειρογνώμονες το λόγο για έναν τελευταίο γύρο παρεμβάσεων, αλλά εφόσον έχουμε χρόνο, διότι δεν έχουμε ε, ερωτήσεις άλλες, βλέπω ότι στο επόμενο σημείο έχουμε το Ρία Ζαχίου από την πρεσβεία της Ινδονησίας που είναι εδώ. Τρία λεπτά σας παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συμφωνήσω με τον πρεσβευτή της Μαλαισίας και ε, να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε το λόγο σε αυτή τη συνεδρίαση. Ε, ε, αναφέρθηκαν κάποιες εξελίξεις στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες ΑΣΕΑΝ και στην Ινδονησία συγκεκριμένα. Πιστεύουμε ότι και η Ινδονησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοούν πολύ καλά την σημασία της πρόθεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη Και της δημοκρατίας. και θέλω να σας αναφέρω κάποιες δραστηριότητες που προσπαθεί η Ινδονησία να προάγει για να βελτιώσει την επαφή της κοινωνίας των πολιτών μεταξύ Ινδονησίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ινδονησία για δεύτερη φορά οργανώνει τις υποτροφίες ε, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν και ε, πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφέραμε πέρυσι μια υποτροφία ε, για συμμετέχοντες στις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και για φίλους της Ευρώπης και για κάποιους που κάνουν ασιατικές σπουδές. Δεύτερη φορά λοιπόν κάνουμε αυτή την υποτροφία, δίνουμε αυτή την υποτροφία φέτος. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα ε, να έρχονται σε επαφή με θρησκευτικούς ηγέτες, με ερευνητές, με ακαδημαϊκούς να συμμετέχουν σε σεμινάρια και έχουν την ευκαιρία να συζητούν με φοιτητές των πανεπιστημίων για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένεσης. Οργανώνονται και επισκέψεις ε, Ινδονησίων ερευνητών από γνωστά πανεπιστήμια, καθώς ε, και ε, από θρησκευτικούς φορείς θα συζητηθεί το θέμα της διαχείρισης της ε, κοινωνικής και θρησκευτικής πολυμορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα ε, των εξτρεμισμών επίσης, ε, γιατί είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν και η Ινδονησία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώνουμε επίσης ένα σεμινάριο ε, για την Ινδονησία που οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ασχολείται και αυτό το σεμινάριο με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω ότι ο κύριος Μαγκόβεν έθιξε και το θέμα ε, της ανεξιθρησκείας στην Ινδονησία. Είναι ένας τομέας στον οποίο μπορούμε να διδαχθούμε ε, ημένα από τους ΔΕ, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και η Ινδονησία. προσπαθούμε να προάγουμε την ε, επαφή μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και να ενισχύσουμε τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ινδονησίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, και πάλι θα ήθελα να σας πω ότι λυπάμαι διότι λόγω εσωτερικών προβλημάτων που είχαμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε από κοινού την τωρινή συνεδρίαση με την συνεδρίαση της αντιπροσωπείας για την Ασία. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Λάγκεν για να δούμε πώς μπορεί να βρεθεί κάποια άλλη λύση για να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Τώρα όμως έχω την κατανόησή σας φαντάζομαι αν σα πω ότι πρέπει να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό θα δώσω το λόγο σε όσους παρενέβησαν ε, και στην αρχή της συνεδρίασης, αν θέλετε το λόγο βέβαια. Ένα θέμα νομίζω ότι αφορούσε την Διεθνή Αμνηστία, οπότε δίνω το λόγο σε εσά, την κυρία Ιζαμπέλ Αχαντών. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εκπροσώπους ε, κυβερνήσεων των χωρών ΑΣΕΑΝ σήμερα στη συνεδρίαση αυτή. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να ακούσουμε και τη δική σας άποψη για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Και θα είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση. και το θέμα της επικύρωσης της ε, Σύμβασης για τους πρόσφυγες ε, που αναφέρθηκε και θέλω να το αναφέρω άλλη μια φορά γιατί η επικύρωση θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία των ε, προσφύγων. Τέλος, είτε μιλάμε για ε, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, είτε ε, για εκπροσώπους κυβερνήσεων, είναι σημαντικό να υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και από νομικής πλευράς και στην πράξη και από όπου και αν προερχόμεθα, γιατί όλοι προερχόμεθα από διαφορετικές κατευθύνσεις, όλοι καλό θα ήταν να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα στην Νότια Ανατολική Ασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ιζαμπέλ. Ο κύριος Μαγκόβεν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ επίσης τους αντιπροσώπους, τα μέλη, πρέσβεις, συμβούλους ε, για τις παρεμβάσεις ε, από πλευρά σας. Πρώτα, ίσως, δύο λόγια για να τονίσω ένα σημείο που αντανακλά, απηχεί ακριβώς αυτή την αυτό το στόχο του να έχουμε υπέρμαχους ε, των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να προαχθεί η επίδοση όσον αφορά τη σημείωση πρόοδου. Ένα από τα πιο σημαντικά σπουδαιότερα βήματα όπως είδαμε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ήταν η απόφαση από πλευρά τη Ινδονησίας και της Ταϊλάνδης να διορίσουν εκπροσώπους ε, της κοινωνίας των, πολιστών, των πολιτών στην ΑΙΤΣΑ. Ένας από τους περιορισμούς ήταν ότι είχαμε εκπροσώπους κυβερνήσεων και όχι τόσο εκπροσώπους ανεξαρτήτων ε, θεσμών και οργάνων. Έκαναν αυτό το βήμα λοιπόν η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία με την επιλογή αυτή της πρωτοβουλίας έχοντας ε, ως δυνατότητα αξιόπιστους έγκριτους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για την παρακολούθηση των θεμάτων των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και θα... είναι μια προοπτική ε, για το μέλλον να υπάρξουν θετικές εξελίξεις περαιτέρω και σε σχέση με την ΑΣΕΑΝ και την Επιτροπή για τις Γυναίκες και τα Παιδιά από την ΑΣΕΑΝ να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχουν σημαντικές επιτροπές για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και εδώ πάλι σε σχέση με την Εθνική Επιτροπή της Ινδονησίας ε, για την προαγωγή των θεμάτων των γυναικών που είναι ένας από τους πιο δυναμικούς θεσμούς και πιο αποτελεσματικούς θεσμούς στην χώρα και στην περιοχή ευρύτερα και ένας από τους σημαντικότερους εταίρους σε σχέση με τα ε, εθνικά θεσμικά όργανα με τα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Για τα δικαιώματα του ανθρώπου, χαίρομαι ιδιαίτερα το ότι αυτό προκλη... ξένησε ενδιαφέρον ε, και προώθησε τη συζήτηση. Και σε σχέση με κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, θα ήθελα να πω ότι θα ήταν χρήσιμο να δούμε κάποια πράγματα. Όπως είπα, τα τέσσερα θεσμικά όργανα από πλευρά ΑΣΕΑΝ έχουν συνενωθεί για να δημιουργηθεί το φόρουμ της Νοτιοανατολικής Ασίας από πλευρά των εθνικών θεσμικών εκπροσώπων και οργάνων. Εργάζονται από κοινού σε κοινά σχέδια και προγράμματα. Ένα από αυτά είναι το εμπόριο, οι επιχειρήσει και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εδώ υπάρχει άμεση παράλληλη διασύνδεση με τα θεσμικά όργανα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση που εργάζονται σε σχέση με την εκπόνηση εθνικών προγραμμάτων δράση θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή εταιρική σχέση ε, μεταξύ των ε, θεσμικών ε, οργάνων εκπροσώπησης των κρατών μελών της ΕΕ και των εταίρων από πλευράς της Νοτιοανατολικής Ασίας για το πώς μπορούν να καταβάλουν από κοινού προσπάθειες να ευδοκιμήσουν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και όπως προανέφερα υπάρχει και το θέμα της εταιρικής ευθύνης. Το θέμα της εταιρικής ευθύνης από πλευράς επιχειρήσεων για αυτά τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Υπάρχουν πλαίσια σε σχέση με τη συμμόρφωση, εκθέσεις για τη συμμόρφωση ε, σε σχέση με αυτές τις προδιαγραφές. Το να συνεισφέρει μια μελέτη που συντάσσεται από το κέντρο των ε, χωρών ΑΣΕΑΝ για τους ανθρώπινους ε, πόρους ε, υπό έναν επαΐοντα που διεξάγει, συντονίζει αυτές τις έρευνες όπου εξετάζεται το πώς εντάσσονται οι αρχές των Ηνωμένων Εθνών σε πολιτικές για, και ένα νομικό πλαίσιο και για τις δράσεις των επιχειρήσεων στην Νοτιοανατολική Ασία. Εκπροσωπούνται λοιπόν εδώ οι προσπάθειες και από πλευράς των κρατών μελών της Νοτιοανατολικής Ασίας και πρότυπα επιχειρησιακά. Είναι μια πολύ καλή θετική συγκυρία να συνδέσουμε και να ανταλλάξουμε πείρα και εμπειρίες με του εταίρους μας της Νοτιοανατολικής Ασίας Εμεί ω Ευρωπαίοι. Είναι ένας τομέα όπου οι Ευρωπαίοι, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν πραγματικά να συνεισφέρουν με μια πρόσθετη ε, αξία που μπορεί να δημιουργηθεί ε, συμμεριζόμενοι εμείς από πλευράς μας ε, την πείρα και την εμπειρία μας με τους εταίρους μας της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε και να υποστηρίξουμε σε τα μάλα αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ all uh, Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους εσάς που συμμετέσχετε ε, σε αυτή τη ε, συζήτηση. Ελπίζουμε ότι αυτές οι συστάσεις θα τηρηθούν και θα δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ε, θα συνεδριάσει το Διευρυμένο Προεδρείο. Θα είναι μια κλειστή συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών που θα ξεκινήσει σε 10 λεπτά περίπου.